da. Da. Hinsetzen. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Wir haben auch heute Καλημέρα αγαπητοί Sinadelfi. Ξεκινάει η σημερινή συνεδρίαση ακριβώς την ώρα της. Ελπίζω να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Ωραία. Η συνεδρίασή μας μεταδίδεται και στο διαδίκτυο, οπότε οι συζητήσεις μας μπορούν μπορεί να τις παρακολουθήσει κάποιος και εκτός της αιθούσης. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, κατά τη διάρκεια του πρωινού 37 φοιτητές του Πανεπιστημίου του Μοντεσκέ από το Μπορντό θα είναι καλεσμένοι μας εδώ πέρα. Θα τους αναγγείλω, μάλλον όταν θα μπουν πάρα πολλοί νεαροί ταυτόχρονα, θα καταλάβετε, αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι, δεν ξέρω μάλλον για, για το μάθημά τους είναι αναγκασμένοι να είναι εδώ, δεν νομίζω να είναι έτσι και ο παδί Ähm, λοιπόν, για να περάσουμε τώρα στην συζήτηση της ε, περιφερειακής ε, διαρθρωτικής ε, πολιτικής και στη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Θα γίνει αυτό με τον γνωστό και καθιερωμένο τρόπο. Ξέρετε, θα δώσουμε πέντε λεπτά στους συγητές για εισαγωγή, μετά θα έχει από 10 λεπτά ο κάθε επίτροπος και μετά θα κάνουμε το γύρο των ομιλητών των ομάδων και κατόπιν είτε πρόεδρος Επιτροπής ε, Περιφερειακών Υποθέσεων ή Κοινωνικών Υποθέσεων, όποιος είναι εδώ πέρα, μετά τους ομιλητές θα λάβει τον λόγο αν το επιθυμεί. Και Κατόπιν θα έχουμε τον πρώτο γύρο των απαντήσεων, αλλά βεβαίως θα παρακαλέσουμε και τους επιτρόπους να είναι σύντομοι, δεν χρειάζονται πολλά λόγια και μετά θα περάσουμε στον δεύτερο γύρο. Σαφές είναι πως ε, καλωσορίζω πρώτα απ' όλα βεβαίως τον Επίτροπο, τον κύριο Χάν. σαφές είναι πως θα καθίσει εδώ πέρα ο κύριος Χάν μέχρι τις 10 και 30 και μετά θα τελειώσει αυτή η συζήτηση γιατί θα πρέπει να φύγει ο κύριος Επίτροπος. Όλες οι υπόλοιπες ε, ανακοινώσεις θα γίνουν μετά, γιατί δεν έχει νόημα τώρα να τρώμε από τον λίγο χρόνο που έχουμε τον κύριο Επίτροπο. Οπότε εγώ θα μείνω μέχρι το τέλος συνεδρίας, μην ανησυχείτε, θα τα πούμε μετά. Οπότε περνάμε στην ε, συζήτηση των ε, περιφερειακών ταμείων και κυρίως το πώς θέλουμε να τα διαμορφώσουμε. Ο Σαλβαδόρ Γκαρίγκα έχει το λόγο για πέντε λεπτά. Gracias, Presidenta. Espero... Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω οι υπόλοιποι συνάδελφοι να μην αντιμετωπίσουν τα τεράστια προβλήματα που αντιμετώπισα εγώ για να καταφράσω στο Κοινοβούλιο γιατί πραγματικά υπάρχει μεγάλη συμφόρηση στους δρόμους και φαντάζομαι πολλοί συνάδελφοι το ίδιο πρόβλημα έχουν γι' αυτό καθυστέρησαν αλλά μια και ο Επίτροπος ε, δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του θα περάσουμε αμέσως στο κυρίως θέμα. Λάβαμε τις απαντήσεις των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων και είναι σαφές από αυτές ότι μια κοινή ανησυχία μας είναι οι δημοσιονομικές περικοπές και η ανάγκη και ο κοινοτικό προϋπολογισμός να υπάγεται στις αρχές της επικουρικότητας και ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας κατά την επιλογή των πολιτικών και των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται φυσικά η πολιτική συνοχής. Κατά τη γνώμη του εισηγητού, και η πολιτική συνοχή αλλά και ο κοινοτικό προπολογισμό δεν θα πρέπει να υποστούν μια γενική μείωση και περικοπή, αλλά να θεωρηθούν ως ε, δραστήρια και αποτελεσματικά όργανα για την επιδίωξη των στόχων της στρατηγικής του 2020 και κυρίως της ανάγκης οικονομικής ανάκαμψης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Γι' αυτό θα έλεγα ότι η περιφερειακή πολιτική δεν είναι κοινωνική πολιτική αμυγός, αλλά ίσως ο πιο αποτελεσματικός οικονομικός παράγοντας για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υλοποιήσει τους στόχους της και να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες των πολιτών της. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον Επίτροπο και να τον ευχαριστήσω για την ε, ροή πληροφοριών που είχαμε τις τελευταίες μέρες. Ποιο θα είναι το μέλλον της πολιτικής συνοχής στο μελλοντικό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πιστεύετε ότι στην πολιτική, περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να έχει ένα τμήμα σε όλες τις πολιτικές ή είναι μια αυτόνομη πολιτική με δική της ξεχωριστή διάρθρωση. Γιατί είδαμε ότι υπάρχουν ανάγκη χρηματοδότησης των νέων πολιτικών, ιδιαίτερα αυτών που απορρέουν από την εφαρμογή της συνθήκης του Λισαβόνας και είδαμε το ρόλο των διαρθρωτικών ταμείων και της περιφερειακής πολιτικής στη χρηματοδότηση αυτή. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε τη γνώμη του Επιτρόπου ποιος θα είναι ο μελλοντικό προσανατολισμός της περιφερειακής πολιτικής. Κάτι άλλο που μας ανησυχεί τα μάλα είναι πώς θα, χρηματοδοτούν, θα χρηματοδοτηθούν οι πιο σημαντικές πρωτοβουλίες, τα flagships που λέμε της πολιτικής της στρατηγικής του 2020, γιατί έχουμε πολλές ανησυχίες ως προς την δημοσιονομική ποσοτικοποίηση, αν θα υπάρχει καταρχήν ή αν αυτές οι ε, πιο σημαντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς θα χρηματοδοτηθούν. Ποια είναι η γνώμη σας. Στο μέλλον, αυτές οι συμβάσεις αναπτυξιακής εταιρικής σχέσης που ήδη εν μέρη άρχισαν να ισχύουν, πώς θα διαμορφωθούν στο μέλλον. Θα τους αποδώσετε ιδιαίτερη σημασία κύριε Επίτροπε, γιατί αυτές οι αναπτυξιακές συμβάσεις μπορούν να βοηθήσουν σε ένα πολύ πιο συνεκτικό προγραμματισμό των ε, μελλοντικών διαρθρωτικών ταμείων και κονδυλίων. Μας ενδιαφέρει να μάθουμε και το επίπεδο στο οποίο θα αναπτυχθούν αυτά, αυτές οι συμβάσεις, αυτά τα μέσα, σε περιφερειακό επίπεδο, σε τοπικό, σε εθνικό. γιατί πολλοί ζητούν να γίνει εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο για να αναμειχθούν όσο, όλο και περισσότερο οι τοπικοί εταίροι, για να αποφύγουμε αποτυχία και τη στρατηγική του 2020 παρόμοια με αυτή που σημειώσαμε στην ε, στρατηγική της Λισαβόνας. Θέλουμε μια περιφερειακή πολιτική φυσικά που θα είναι προσανατολισμένη σε αποτελέσματα, βελτίωση του συντονισμού μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών. Εμείς Πιστεύουμε στην αρχή της συγκέντρωσης και θέλουμε να μας πείτε και τη γνώμη σας. Και ως προς την αιρεσιμότητα, δεν είναι ακόμη σαφές στην Επιτροπή μας ποια θα είναι τα κριτήρια, τα πιο προνομιακά κριτήρια αιρεσιμότητας για την εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά το σύμφωνο σταθερότητας, αλλά και την ε, υλοποίηση των στόχων που προσδιορίζονται σε αυτές τις ε, αναπτυξιακές συμβάσεις. Αυτά κύριε Πρόεδρε και περιμένω τις παρατηρήσεις και των λοιπόν συναδέλφων που φαντάζομαι θα είναι εύστοχες και πιο συγκεκριμένες από τις δικές μου. Ε. ναι, ευχαριστώ πολύ. Τέλεια προς το χρόνο. Οπότε τον λόγο έχει ο κύριος Επίτροπος για 10 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο εισηγητή, ο οποίος ανέφερε τα βασικότερα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως η περιφερειακή πολιτική είναι μια εγκάρσια πολιτική η οποία οδηγεί με ολοκληρωμένο τρόπο στην ανάπτυξη των περιφερειών και συνολικά των κρατών μελών. Η πολιτική συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία είναι όπως ε, είπε στο έγγραφο εργασία υπαριθμών 2 και αναφέρω ακριβώ. παίζει ρόλο κλειδί όσον αφορά τι προτεραιότητε μια έξυπνη και αηφόρου ανάπτυξης στα κράτη-μέλη και τις ε, περιφέρειες και θα πρέπει να διαμορφωθεί ως δυνατόν πιο αποτελεσματικά για να ενισχύσουμε περισσότερο στόχους Ευρώπης 2020. Βρισκόμαστε τώρα στο δεύτερο μισό της ε, προγραμματικής οικονομικής περίοδου και μπορώ να σας πω πως ε, τα προγράμματα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Βεβαίως ε, βλέπουμε πως κάποια δεν είναι σε... Κατηγορούνται ορισμένα κρατημέλη ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν πλήρως τα διαρθρωτικά ταμεία, κάτι το οποίο είναι λανθασμένο και φαίνεται αυτό σε κάποια διαγράμματα για την πολιτική συνοχή. Σε έφερα μαζί σας ε, κάποια φύλλα, δεν μπορείτε να τα δείτε από τη θέση μου. Τέλος πάντων θα σας τα πω με λόγια. Το απλό έχουμε προγραμματικούς κύκλους στις ε, διάφορες ε, περιόδους οι οποίοι οδηγούν σε κάποιες αλληλεπικαλύψεις. Αν έχουμε μία περίοδο ε, όπως από το 2000 μέχρι το 2006 οι τελευταίες πληρωμές πάνε μέχρι το έτος 2012. Το ε, επόμενο έτος δηλαδή. Και βεβαίως ε, οι πληρωμές για την τρέχουσα περίοδο έχουν ήδη ξεκινήσει. Οπότε βλέπετε εδώ πέρα, δεν ξέρω αν βλέπετε αυτές τις στήλες από μακριά, την χρήση των ε, κρατών μελών ε, στα διάφορα έτη, στα η οποία παραμένει λίγο πολύ σταθερή ανεξαρτήτως του εάν μιλάμε για τα παλιά ή τα νέα προγράμματα. Έτσι, παραδείγματο χάρη, το 2010 μόνο από τον τομέα της ε, DG Regio μιλάμε για πάνω από 30 δισεκατομμύρια σε πληρωμές, ενώ το 2008 είχαμε μια αύξηση σε σχέση με το 2008 κατά 10% κατά το οποίο είναι απολύτως συγκρίσιμο με τις φάσεις στην προηγούμενη περίοδο. Η περιφερειακή πολιτική δρά στο επίπεδο της περιφερειακής οικονομίας και βλέπετε πως από το 2000-2006 δημιουργήθηκαν γύρω στο 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας και το ΑΕΠ στις περιοχές στόχου 1 αυξήθηκε 10 με 15% και διάφορες μελέτες αποδεικνύουν πως και στις χώρες οι οποίες είναι καθαροί εισφορείς οδηγεί σε αύξηση των εξαγωγών και του ΑΕΠ, κάτι το οποίο βοηθά βεβαίως στην εξίσωση των πληρωμών αυτών. Διάφορα μοντέλα μακροοικονομικής πολιτικής δείχνουν πως η πολιτική συνοχής συνολικά, εάν κάνουμε έναν απολογισμό, έχει αυξήσει το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε μπορούμε να την αντιληφθούμε ως μια πολιτική επενδύσεων. Αλλά βεβαίως υπάρχει και η διάσταση της αλληλεγγύης. Αλλά η πολιτική συνοχής δεν μπορούμε να την δούμε ως μόνο μια πολιτική συνοχής ή πολιτική αλληλεγγύης. Και οι δύο διαστάσεις ισχύουν. Η περιφερειακή πολιτική επίσης δεν μειώνεται μόνο στα θέματα από τα οποία αποτελείται. Αποτελεί θα έλεγα θεμέλιο λίθο για μια έξυπνη και αηφόρο ανάπτυξη και η περιφερειακή πολιτική ούτως ή άλλως έχει έναν έξυπνο αηφόρο και κοινωνικά ενταξιακό χαρακτήρα προέρχεστε όλοι από κάποιες περιφέρειες και ξέρετε πόσο διαφορετικές είναι μεταξύ τους. Η πολιτική συνοχής πρέπει και αυτό κάνει βεβαίως να λαμβάνει υπόψη όλες τις πτυχές ε, Τη πολιτική επενδύουμε ήδη σε αυτή την περίοδο πάνω από 500 δισεκατομμύρια ε, ευρώ στην ε, αηφόρο ανάπτυξη και 86 δισεκατομμύρια στην έρευνα και ανάπτυξη και στην καινοτομία περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πολιτική της Ένωσης και βεβαίως αυτό φαίνεται και στην δομή του προϋπολογισμού και εδώ πέρα συμφωνώ με την ε, άποψη και τις αμφιβολίες ε, της κυρίας Γκρέλ στην τοποθέτηση Επιτροπής Περιφερειακών Θεμάτων πως δεν θα είχε νόημα να πάνε σε διαφορετικά κεφάλαια του προϋπολογισμού τα διαρθρωτικά ταμεία και να διακινδυνεύσουμε έτσι την ενότητα αυτό ακριβώς είναι προς το συμφέρον ε, των ε, κρατών και των περιφερειών για να μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα σε περίοδους κρίσης. Όμως αυτό σημαίνει πως πρέπει να εξελιχθούμε γρήγορα, να αντιδρούμε γρήγορα και να αναγνωρίσουμε τα σημεία των καιρών. Έτσι, στην πέμπτη έκθεση την ε, πέμπτη σχετική έκθεση. Έτσι και εγώ και οι συνάδελφοι χαιρόμαστε για το ότι βρήκαμε ισορροπία μεταξύ των αναγκών των ε, περιφερειών και των κρατών. Αν τώρα κάποια ουσιαστικά σημεία τα οποία ανέφερε ήδη εν μέρη ο κύριος συγητής και θα έχουν ε, κάποιες επιπτώσεις στις δημοσιονομικές προοπτικές. Από τη μία υπάρχουν οι πάρα πολλές επιθυμίες και προσδοκίες από την περιφερειακή πολιτική και για να μπορέσουμε να τις προσεγγίσουμε θα έλεγα πως χρειαζόμασταν έναν προϋπολογισμό ο οποίος σε απόλυτα νούμερα είναι λίγο πολύ ε, αυτός που έχουμε. Η ενότητα το δεύτερο κομμάτι πρέπει να ε, παραμείνει κάτι το εγγυημένο. Θα πρέπει να έχουμε δηλαδή ένα κοινό περιφερειακό ταμείο με κοινού κανόνες και αυτό συνεισφέρει στην περαιτέρω απλοποίηση. Ως προς αυτό έκαναν την δουλειά τους οι προκάτοχοί μου και σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο ο αριθμός των διαφόρων προγραμμάτων μειώθηκε και θεωρώ πως αυτό έχει αποδείξει την αξία του στην πράξη. Χρειαζόμαστε ένα απλό σύστημα προωτήσεων το οποίο θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στον δικαιούχο. Αλλά πάντα υπάρχει βεβαίως περιθώριο βελτίωσης, οπότε μιλάμε για ένα έργο σε εξέλιξη απευθύνω έκκληση στα κράτη-μέλη και τις ε, περιφέρειες γιατί κάποια γραφειοκρατία είναι επιπρόσθετη γραφειοκρατία η οποία προστίθεται, αν θέλετε, σωρεύεται πάνω στη δική μας. Καταθέσαμε λοιπόν μια πρόταση για τη μελλοντική πολιτική συνοχή που στοχεύει στο να επικεντρωθούμε στόχους της Ευρώπης 2020 για να έχουμε την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Έχουμε τους όρους ex ante, η οποία μπορεί να συμφωνηθεί μόνο με τα κράτη-μέλη και η οποία θα ε, εγγυηθεί πως οποιοδήποτε αιτία που γνωρίζουμε σήμερα ότι οδηγεί σε καθυστέρηση εφαρμογή των έργων στις διάφορες περιφέρειες και χώρες να αντιμετωπιστεί από κοινού με τα κράτη-μέλη. Γρήγορα και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις ε, στην εφαρμογή. Για αυτή την αιρεσιμότητα και τα διάφορα παραδείγματα Ξέρετε πως αυτά μπορούμε να τα συμφωνήσουμε μόνο από κοινού με τα κατημέλη και αποτελούν ένα παράγοντα επιτυχίας. Επίσης προβλέπουμε πως θα έχουμε δείκτες αποτελεσμάτων που θα οριστούν σε συμφωνία με τα κράτη-μέλη και θα υπάρχει και το ζήτημα της αναλογικότητας το οποίο θα λάβουμε υπόψη. Οπωσδήποτε θα ρωτήσετε τι θεωρώ για την χρονική διάρκεια του προγράμματος πλαισίου. Κοιτάξτε, λιγότερο από 7 χρόνια δεδομένη της φύσης των έργων μας ε, την θεωρώ μια προβληματική περίοδο. Συμπεράσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μετά την ε, τελευταία οικονομική κρίση ενώπιον τεράστιων προκλήσεων. Από την άλλη πρέπει να δούμε θα κάνουμε με τον προϋπολογισμό, αλλά αντιστρόφως και να φροντίσουμε την ανταγωνιστικότητα και εδώ πέρα ακριβώς είναι τομέας που θα δράσει η περιφερειακή πολιτική. Θα συνεισφέρουμε με τρόπο ποιοτικό και ποσοτικό στην αναπτυξιακή πολιτική των περιφερειών, όπου με βάση λιγότερων ε, προτεραιοτήτων θα έχουμε λύσεις οι οποίες θα δημιουργηθούν και γι' αυτό χρειαζόμαστε την πολιτική συνοχή και είμαι πεπισμένος ότι χρειαζόμαστε μια πολιτική οποία θα είναι σε θέση να συμβάσει στρατηγική της Ευρώπης 2020 που αυτή τη στιγμή είναι μόνο στα χαρτιά να τη μεταφράσει σε συγκεκριμένες δράσεις και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που τελικά θα συμπεριλάβει περιφέρειες και κράτη-μέλη και μια τελευταία παρατήρηση για να απαντήσω στο ερώτημα του κυρίου συγητή. Θα προβλέψουμε και θα πιέσουμε τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο μιας πραγματικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης ε, να εμπλέξουμε εκ των προτέρων στις ε, διαπραγματεύσεις ε, περιφέρειες στα επιχειρησιακά προγράμματα και στις συμβάσεις εταιρικής σχέσης για να θεωρούν πως πράγματι αυτά τα πράγματα τους ανήκουν και να συνεισφέρουμε σε ότι η πολιτική συνοχής θα είναι μια διαρκής επιτυχία και θα συνεισφέρει στην επιτεύξη των στόχων του 2020. Σας ευχαριστώ. Παραμένετε πιστός ε, στην προσέγγιση της ε, Κομισιόν. Όλοι οι προκατοχοί σας είχαν πει πως ε, η περιφερειακή πολιτική δεν είναι ένα ρημουλκούμενο αν θέλετε, είναι ο κινητήρας της ανάπτυξης και έτσι θα πρέπει να το βλέπουμε. Τώρα ε, θα μιλήσουν των ομάδων για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Τέσσερα λεπτά. Ο Ιαν Ολμπριχτ. <coughs> Κύριε Επιτρόπε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σε όλα τα έγγραφά του διατρανώνει ότι η θεμελιώδης πρόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Γι' αυτό και η πολιτική συνοχής είναι μια πολιτική επενδυτική κατά κάποιο τρόπο και βελτιώνει τις ευκαιρίες για αποκατάσταση των ανισορροπιών στην ανταγωνιστικότητα μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών περιφερειών. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις ως προς το θέμα αυτό, κύριε Επίτροπε. Αν υποθέσουμε ότι η στρατηγική του 2020 δεν ξεκινήσει το 2014, αλλά έχει ήδη αρχίσει το 2010. Αυτό σημαίνει ότι η στρατηγική του 2020 υλοποιείται με τα μέσα και δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια των νέων μέσων. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Επίτροπε, μήπως μετά το 2004 είναι σκόπιμα να τροποποιήσουμε τα μέσα μας. Δηλαδή να τροποποιήσουμε τη δομή των, του προϋπολογισμού εν μέσω της στρατηγικής. Ή ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο τους στόχους. Πώς θα ερμηνεύσουμε εμείς. Γιατί το αναφέρατε κι εσείς, ε, κύριε Επίτροπε, για τα θέματα της συνοχής. τις διάφορες διαστάσεις πώς θα τις αντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο της ε, ε, πολιτικής συνοχής και ποια η σχέση αυτής με τις εμβληματικές πρωτοβουλίες. Γιατί έχουμε μια ολόκληρη διαδικασία που ήδη έχει ξεκινήσει. Ερωτώ λοιπόν, σε ποιο βαθμό θέλουμε να υλοποιήσουμε τα συγκεκριμένα στοιχεία. Δεύτερον, πιστεύετε κύριε Επίτροπε ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στον τρόπο εφαρμόγης αυτής της πολιτικής. Γιατί είναι σημαντικό αυτό για τον προϋπολογισμό, γιατί εμπίπτει στην αρχή του short management. Επίσης, μια και εμπίπτει σε αυτή την κοινή διαχείριση, το shared management, και επειδή είπαμε ότι θα πρέπει να δώσουμε και πολυεπίπεδη διάσταση, πώς θα υλοποιήσουμε αυτή την πολυεπίπεδη διάσταση και την ε, κοινή διαχείριση και πώς αυτό θα το αντιμετωπίσουμε σε διάφορες συμβάσεις αναπτυξιακής εταιρικής σχέσης. Και σε ό,τι αφορά το εύρο ε, των οικονομικών, αν υποθέσουμε ότι δεν θα αλλάξουν οι αναλογίε του προπολογισμού και τα κονδύλια θα μείνουν τα ίδια, αυτό σημαίνει ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να καλύψει όλε τι περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το λογικό συμπέρασμα. Οπότε η πρότασή σα, κύριε Επίτροπε, είναι μια πολιτική που δεν αφορά μόνο τις αδύναμες περιοχές, αλλά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επικράτησης. Θα γίνει κάποια αλλαγή ως προς αυτό. Γιατί αν ε, γίνουν τέτοιες αλλαγές, ε, θα είναι τεράστιες ε, οι επιπτώσεις για το εύρος της πολιτικής συνοχής. Εμείς, το ΕΛΚ, Είμαστε υπέρ της α, σημερινής, του σημερινού των οικονομικών, αλλά θέλαμε να μάθουμε και τη δική σας γνώμη ως προς τις διαστάσεις αυτές. Ευχαριστώ. Γιάν, η επόμενη ομιλήτρια είναι η Κωνσταντσε για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Να ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω τη σημασία της ε, περιφερειακής ε, πολιτικής και της πολιτικής συνοχής. Απλά σημαντικό για εμάς είναι πως η πολιτική συνοχής δεν είναι μόνο μια οικονομική πολιτική, είναι μια πολιτική της συνοχής όπως λέει και η λέξη. Γι' αυτό πρέπει να συμμετέχουν όλες οι περιφέρειες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ακούσαμε πως προτείνουν μια τέτοια κατανομή για την πρόσβαση στα μέσα συνοχής της Ένωση. Για εμά είναι σαφέ πω πρέπει να έχουμε προτεραιότητες. Ίσως λοιπόν ο κύριος Επίτροπο μπορεί να μας εξηγήσει ποιε προτεραιότητε θέλει να προτείνει για να δημιουργηθεί ακριβώ μια τέτοια συνοχή σε ολόκληρη την Ένωση. Είμαστε σε δύσκολες ε, συνθήκες ε, οικονομικές και γνωρίζουμε τι γίνεται με τον προϋπολογισμό των κρατών μελών. Γι' αυτό είναι σαφές πως θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τα μέσα στην ε, διάθεσή μας και βεβαίως παρά το ότι η Κομισιόν και, η κράτη και τα κράτη-μέλη εργάζονται σε αυτό, εξακολουθούμε να έχουμε έλλειμμα στην αποτελεσματική χρήση των πόρων. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, να είναι η έλεγχη διαφανή αλλά όχι υπερβολικά γραφειοκρατική. Μπορεί να μας πει λοιπόν ο κύριος Επίτροπος τι σκοπεύει να κάνει για την μελλοντική προγραμματική περίοδο και ποια πράγματα προτείνει. Και ίσως να μας πει τι σημαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή προσανατολισμένο στα αποτελέσματα. Θα θέλαμε να μας πει πώς θα εφαρμοστεί. Τώρα όταν μιλάμε για αποτελεσματική χρήση των πόρων, νομίζω πως εκεί πέρα ε, πρέπει να δούμε και τον συντονισμό. Ίσως θα μπορούσαμε λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε πως τι θα γίνει με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην ε, πολιτική συνοχής και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς τι γίνεται με την αγροτική ανάπτυξη με το Γεωργικό Ταμείο εκεί πέρα και ποιες ιδέες έχει σχετικά η Κομισιόν. Μας ενδιαφέρει λοιπόν πάρα πολύ αυτό και σε μια προηγούμενη συνεδρίασή μας ακούσαμε διαφόρους επιτρόπους ε, που μίλησαν για ταμεία, για το πώς θα βρουν λεφτά, όχι μέσω της αύξησης του προϋπολογισμού της Ένωσης, κάτι το οποίο είναι δύσκολο, αλλά σκέφτονται την πολιτική συνοχής που θα τα χρηματοδοτήσει όλα αυτά. Όμως επειδή η πολιτική συνοχής δεν είναι μόνο πολιτική συγκοινωνιών ή ε, μόνο πολιτική έρευνα ή μόνο ενεργειακή πολιτική, τι άποψη έχει ο κύριος Επίτροπος για τα νέα ταμεία ή για το να χρησιμοποιηθεί ε, η πολιτική συνοχής για άλλους τομείς πολιτικής ε, της Ένωσης. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Επίτροπε. Μιλάτε για έξυπνη προσέγγιση, ναι. Αλλά πώς θέλει να κάνει κάτι τέτοιο η Κομισιόν, γιατί μέχρι στιγμής δεν βλέπω να έχει υπάρξει κάποια πρόοδος ή διαπραγμάτευση με απευθείας με τις περιφέρειες και θα ήθελα μια απάντηση εδώ πέρα και τι άποψη έχει η Κομισιόν για τα μη διατεθέντα κονδύλια τα οποία θα έπρεπε να επιστρέφουν στην Κομισιόν και όχι στα κράτη-μέλη. Εμεί θα δώσουμε τη μάχη ως Κοινοβούλιο, αλλά τι μπορεί να κάνει και η Κομισιόν για να μας βοηθήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια χαρά όσον αφορά το χρόνο. Ναι, πρέπει, πρέπει να είμαι αυστηρή, αλλιώ ε, θα μιλήσουν λίγοι. Οπότε Όταν λέω τέσσερα λεπτά, δεν ανάγκη να τα εξαντλήσετε και τα τέσσερα και λιγότερα γίνεται. Για το Άλντε λοιπόν. Thank you, Mrs. Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε για την καλή σας παρουσίαση. Η πολιτική συνοχής πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Ε, επιφέρει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και είναι στο επίκεντρο της ε, Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2020. Χωρίς μια ευρεία και δυνατή περιφερειακή πολιτική δεν μπορούμε να έχουμε ενέργεια, καινοτομία που να είναι δυνατές. Επίσης θα πρέπει στην πολιτική συνοχή να κάνουμε κάποιες αλλαγές και η ομάδα μας το πιστεύει αυτό. Χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικές πολιτικές που να συνδέονται με τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Νομίζουμε ότι η έκθεση για τη συνοχή λοιπόν ήταν μια καλή εκκίνηση. Το νέο, ε, νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, θα πρέπει να συνδέσει διάφορα στοιχεία πιο έντονα μεταξύ τους. Η πολιτική συνοχής ε, ήταν και στο παρελθόν ε, σημαντική γιατί υλοποίησε την ε, πολιτική ε, της Λισαβόνας. Θα πρέπει να βρει τώρα και τα κονδύλια για να υλοποιηθεί η στρατηγική 2020 στη Λισαβόνα. Στα πλαίσια της Λισαβόνας χρειαζόμαστε αυτά τα κονδύλια για τους 15 της Ευρώπης. Το 60% των κονδυλίων ε, πηγαίναν στην, ε, για τη στρατηγική της Λισαβόνας και το 75% για, την, ε, για το, την περιφερειακή ανάπτυξη. και πρέπει να παραδεχθούμε ότι ορισμένες περιοχές που το χρειάζονταν πήραν 90% των κονδυλίων. Θα πρέπει να το εξασφαλίσουμε και στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Τώρα για τις καινοτομίες θα πρέπει να τη συνδέσουμε ακόμη περισσότερο με την πολιτική συνοχή, ε, συνοχής. Το 5% της καινοτομίας συμβαίνει στην ε, τεχνολογία και στην επιστήμη, σε αυτούς τους τομείς. Δεν θέλω να τα υποτιμήσω αυτά, αλλά το 95% σχεδόν 100 των καινοτομιών είναι ε, πολύ συγκεκριμένα πράγματα ε, και έχουν, ε, προωθούν μια σχέση πελάτη εταιρεία. Επομένως, η πολιτική συνοχή θα πρέπει να παίξει το ρόλο της για να επιταχυνθεί η καινοτομία. Και φυσικά πολλές από αυτές τις γνώσεις υπάρχουν στις περιφέρειες. Οι περιφέρειες μπορούν να παίξουν λοιπόν το ρόλο τους. Κύριε Επίτροπε, αυτές τις προκλήσεις πώς μπορεί να τις αντιμετωπίσει η πολιτική συνοχής. Ε, πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτές τις πολύ συγκεκριμένες καινοτομίες στα πλαίσια της έρευνας και της τεχνολογίας. Στα, στους διάφορους τομείς της ε, πολιτικής συνοχής η εδαφική συνεργασία είναι πολύ σημαντική. Έχουμε τις μακροστρατηγικές, χρειαζόμαστε και σαφή σχέδια. Τι, σχέδια έχετε εκπονήσει κύριε Επίτροπε για αυτές τις στρατηγικές, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά. Χρειαζόμαστε μια πανευρωπαϊκή πολιτική συνοχής. Και νομίζω ότι χάρη σε αυτό μπορούμε να υλοποιήσουμε και τους στόχους ε, της Ευρώπης 2020. Ευχαριστώ τώρα για τους πράσινους, Φρανσουά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για μας η πολιτική συνοχής είναι η ψυχή της ευρωπαϊκής πολιτικής. Κάθε λαός και κάθε έδαφος νομίζω εκεί προωθεί την, ε, και προβάλλει τις ελπίδες του. Και επομένως ε, για μας χρειάζεται μια βιώσιμη πολιτική συνοχής που να εγγράφεται σε ένα μακροχρόνιο ορίζοντα. Η σημερινή περίοδος προγραμματισμού ε, χαρακτηρίστηκε από ένα ιστορικό γεγονός, ε, η ένταξη των 10 νέων χωρών με μεγάλη καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους. Ε, δεν θα πρέπει να μείνουμε εδώ τώρα. Θα πρέπει να εμπνευστούμε και να φτιάξουμε μια νέα αρχιτεκτονική. Αυτό το απαιτεί και η συνθήκη της Λισαβόνας, γιατί η εδαφική συνοχή σήμερα είναι υποχρέωση της ε, Ένωσης. Ε, όλοι πρέπει να ασχοληθούμε και κυρίως ε, και οι Κομισιόν με βάση τις συνθήκες. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσει μια πολιτική συνοχής με διάρκεια ούτως ώστε ο μηχανισμός ο οποίος υπήρχε μέχρι σήμερα να αναπροσαρμοστεί. Ο Επίτροπος ανέφερε κάποια πράγματα, αλλά δεν μας ικανοποιούν όλα. Άλλα μας ικανοποιούν και άλλα μας φαίνονται ανεπαρκή. Ε, κάτι το οποίο κατά την άποψή μου πήγαινε προς σωστή κατεύθυνση είναι η, ε, η δημιουργία ενός ενδιάμεσου στόχου μεταξύ του 1 και του 2. Αυτό μου αρέσει και μας επιτρέπει να καθορίσουμε ένα στόχο μακροπρόθεσμο για την πολιτική συνοχής το 75% είναι ένας στόχος σημερινός σε σχέση με τις καθυστερημένες περιοχές, ε, οι οποίες θα πρέπει να είναι προτεραιότητα, ούτω ώστε η κάθε περιοχή να ξεπεράσει τα σημερινά της ε, εμπόδια. Για μας όμως πρέπει να πάμε ακόμα πιο μακριά. Πρέπει σε αυτή την πολιτική συνοχής να δώσουμε ένα μακροπρόθεσμο στόχο, συγγνώμη, σύμμορφο με τις ανάγκες ε, που αντιμετωπίζουμε. Σήμερα υπάρχει οικονομική κρίση μπροστά μας, η οποία πιέζει αρνητικά τις ε, φιλοδοξίες της μελλοντικής πολιτικής συνοχής. Ε, εσείς θέλετε να διατηρήσετε το δημοσιονομικό φάκελο αυτό και τα κονδύλια για την πολιτική σας, αλλά βλέπω τα, μηχανάκια του, τους υπολογιστές στα διάφορα Υπουργεία Οικονομικών που θέλουν να σας συμπιέσουν αυτά τα ποσά. Ακόμα και στους διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα ακούμε αυτά. Αυτό είναι κρίμα, γιατί η, κρίση σήμερα δείχνει ότι πρέπει να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε την πολιτική συνοχή. Είμαστε σε φάση δημιουργίας, έτσι λίγο βιαστικά ας πούμε, κάποιους μηχανισμούς για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης αυτό συνδέεται και με τα οικονομικά κυκλώματα της ε, ενίας αγοράς. Πρέπει να δώσουμε ένα αντιστάθμισμα στην ενία αγορά. Και αυτό είναι η πολιτική συνοχής. Για μας είναι πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να την δημιουργήσουμε έτσι βιαστικά, αλλά θα πρέπει να έχει μια διάρκεια. Και αυτή η πολιτική συνοχής ε, κινδυνεύει σήμερα, γιατί θέλουμε να μειώσουμε τις πιστώσεις, ε, όλοι το λένε από διάφορες πηγές, ακόμη και εδώ στο Κοινοβούλιο. Η Ευρώπη θα πρέπει να δώσει τα κονδύλια, ούτω ώστε να υπάρξει ανάπτυξη δίκαιη σε όλη την επικράτειά της και όχι μόνο στις ζώνες που είναι οικονομικά ανεπτυγμένες. Θα πρέπει να υπάρξει επίσης και εδαφική ισορροπία, να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο, ούτως ώστε να βοηθήσουμε τις ε, ε, περιφέρειες που είναι πάρα πολύ πολυπληθείς και να προωθήσουμε τις περιφέρειες οι οποίες δεν έχουν ε, αρκετή πυκνότητα πληθυσμού. Ε, αυτά λοιπόν κύριε Πίτροπε, εμείς θα σας υποστηρίξουμε στην προσπάθειά σας αυτή. Ευχαριστώ. Νομίζω πως ε, μέχρι στιγμής άκουσα πως μόνο ο Γάλλος Υπουργός ε, Οικονομικών ε, θέλει να διαγράψει την πολιτική συνοχή κανέναν, από κανέναν άλλον. Αλλά είναι σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να το δούμε. Τώρα για τους Ευρωπαίους συντηρητικούς ο Ρίτσαρντ Ασχουρθ. Θέλω να κάνω τρεις ερωτήσεις. Ποιος είναι ο στόχος της ε, χρηματοδότησης και των δαπανών. Υπάρχει ε, δεύτερον, υπάρχει προστιθέμενη αξία και δεύτερον, ε, υπάρχει τι παίρνουμε για τα λεφτά που δίνουμε. για την πολιτική συνοχή, η απάντηση στις τρεις ερωτήσεις δεν ξέρω ποια είναι. Δεν είναι σίγουρος ότι είναι θετική. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει οι οικονομικοί πόροι να πάνε με σκοπό την υλοποίηση της οικονομικής σύγκλησης. Νομίζω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον και των πλούσιων και των φτωχών και των ανεπτυγμένων και των μη ανεπτυγμένων χωρών. Αλλά δεν ξέρουμε αν τα σημερινά προγράμματα πραγματικά ε, δίνουν κάτι για τα χρήματα των φορολογουμένων που ξοδεύουμε. Η στρατηγική 2020 θα πρέπει να είναι ο κροκονιαίος λίθος της πολιτικής συνοχής και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και δεξιότητες για τους εργαζόμενους. Η ανάπτυξη των μια μικρή πράσινη οικονομία είναι επιθυμητή και σε αυτού του δύσκολου καιρού είναι μεγάλη ευκαιρία για όλα τα κράτη-μέλη τη Ένωση. Αλλά θα πρέπει να γίνει πειθαρχημένα. Και αυτό τι σημαίνει. Τα κοινοτικά κονδύλια δίδονται σε εκείνε τι περιοχές όπου τα, ε, τα κράτη δεν μπορούν από μόνα του να αναπτύξουν αυτέ τι περιοχέ και η χρηματοδότηση θα πρέπει να δοθεί ούτω ώστε να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δεν θα μπορούσαν αλλιώ να ελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια. Θα θέλαμε σε αυτή την περίπτωση να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα και στην ανάπτυξη, αλλά τονίζουμε ότι αυτή η χρηματοδότηση θα πρέπει να δοθεί με βάση την αριστεία και όχι με κυκλική χρηματοδότηση. Θα πρέπει να υπάρξουν νέε μορφέ ενέργεια ε, χάρη σε αυτά τα κονδύλια και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα, ειδικά με διασυνοριακά δίκτυα ε, και ε, ευρυζωνική σύνδεση. θέλουμε λοιπόν μια, κάποιες υποδομές να προωθηθούν, που υποδομές που στο παρελθόν δεν είχαν πετύχει. θέλουμε επίσης να δοθούν περισσότεροι πόροι στην ενιαία αγορά. Ε, να διευρυνθεί ενδεχομένω, ίσω στον τομέα των υπηρεσιών, η εμβέλεια τη ε, νέα αγορά. Ε, επένδυση στι νέε τεχνολογίε, προγράμματα κρατικών προμηθειών και ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ούτω ώστε να έχουν πρόσβαση στην ενιαία αγορά. Αυτό είναι ένα καλό τρόπο για να ενθαρρύνουμε την οικονομική ανάπτυξη. Τώρα, τέσσερι αδυναμίε. Όπω είπα και πριν, ιστορικά η Κομισιόν στάθηκε αδύναμη στο στην κατηγοριοποίηση των στόχων. Ε, δηλαδή, δεν υπήρχε σωστή ε, αξιοποίηση της χρηματοδότησης, επομένως δεν ε, δόθηκαν σωστά τα χρήματα, ειδικά σε μεγάλα προγράμματα υποδομών. Τα προγράμματα δεν ήταν πολύ αποδοτικά επίσης. Το ελεκτικό συνέδριο ε, ήταν πολύ επικριτικό, ας πούμε, και βρήκε σφάλματα. Η προσέγγιση α, των 27 κρατών επίσης είναι πολύ διαφορετική. Γενικά, ε, είναι εθνικό και πολιτιστικό θέμα. Κάποια κράτη όμως είναι πιο επιχειρηματικά και επομένως έχουν κλίμα έτσι, φιλικό προς επιχειρήσεις, ενώ άλλα όχι. Τώρα, ίσως εκεί και είναι η ώρα, ε, να ανοίξουμε στην επιχειρηματικότητα. Αυτό βέβαια έχει, ε, επηρεάζει την πολιτική συνοχής. Γιατί τελικά αυτά τα κονδύλια τα χρειάζονται οι πιο φτωχέ ε, περιφέρειε και έχουν τη λιγότερη δυνατότητα να απορροφήσουν αυτά τα κονδύλια συνοχή και αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τέλο, είναι σημαντικό τα κονδύλια τη ε, πολιτική συνοχή να μην αντικαθιστά ε, κονδύλια εθνικά. Υποκαθιστά μάλλον κονδύλια εθνικά. Θα πρέπει δηλαδή παρόλα αυτά οι εθνικές χώρες μειώνοντα του φορολογικού συντερεστέ κτλ. Και, και δίνοντα διάφορα κίνητρα, να μπορούν παρόλα αυτά να δίνουν και αυτέ κονδύλια. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε δηλαδή με αυτά τα κονδύλια μια μοντέρνα ανταγωνιστική καινοτομία, ε, τεχνολογίε νέα γενιά, ε, καινοτόμου τρόπου επίση για να δημιουργήσουμε ε, περισσότερε θέσει απασχόληση στα πλαίσια τη στρατηγική 2020 ξεπέρασε το χρόνο κατά 30 δευτερόλεπτα. Εν πάση περιπτώσει. Μιγγέλ Πόρτας τώρα για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Εγώ θα ξεκινήσω την πρώτη μου ερώτηση με ακριβώς αντίθετο τρόπο από αυτό που τελείωσε ο προλαλής σα. Το Ταμείο Συνοχής είναι ένα ταμείο που υπάγεται στην αιρεσιμότητα. Δηλαδή εξαρτάται από το κατά πόσο τα κράτη-μέλη υλοποιούν τα προγράμματά τους σταθερότητα και σύγκληση. Δηλαδή τα προγράμματα λιτότητά του. Από αυτό εξαρτάται αν θα λάβουν τα κονδύλια της συνοχής. Όμως, εν μέσω οικονομικής κρίσης, πώς είναι δυνατόν να ισχυριζόμαστε ότι τα κοινοτικά κονδύλια που είναι απολύτως απαραίτητα για τη συγχρηματοδότηση στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίσουν περισσότερες δημοσιονομικές δυσκολίες, πώς είναι δυνατόν τα κονδύλια αυτά να υπόκειται στην προϋπόθεση τήρησης ε, των ε, προγραμμάτων λιτότητας. Και σε περίπτωση που το, έλλειμμα, το δημοσιονομικό έλλειμμα των κρατών ξεπερνά το 3% δεν μπορούν να λαμβάνουν αυτά τα κονδύλια. Από που ισχύει αυτή η αιρεσιμότητα των ε, κονδυλίων συνοχής μας οδηγεί την παράδοξη κατάσταση οι χώρες που χρειάζονται απολύτως τη χρηματοδότηση για να πραγματοποιήσουν κρατικές επενδύσεις σε μια στιγμή που οι ιδιωτικές επενδύσεις ε, έχουν ε, καταβαραθρωθεί, πώς είναι δυνατόν να επιδιώκεται ανάκαμψη της οικονομίας εφαρμόζοντας τέτοιες προϋποθέσεις. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι η εξής. Στις ε, μίζωνες επενδύσεις υποδομών, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Επίτροπος, θα υπέρ της σύμπραξης ε, ιδιωτικών και κρατικών κονδυλίων. Δηλαδή, θέλουμε να εισαγάγουμε ιδιωτικά κονδύλια υποκαθιστώντας τα κρατικά, αλλά λέμε ότι μέσα σε 20-30 χρόνια το χρέος ε, θα αυξηθεί. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν κύριε Επίτροπε, από τη μία να υποστηρίζουμε μια πολιτική συγκράτηση του δημόσιου χρέους και απ' την άλλη να εφαρμόζουμε μια επενδυτική στρατηγική που θα στηρίζεται σε συμπράξεις ε, κρατικών και ιδιωτικών ε, κεφαλαίων. Η τρίτη μου ερώτηση αφορά την κατάσταση στην Πορτογαλία, την πατρίδα μου. Μία από τις χώρες που υποφελήθηκαν περισσότερο από τα κονδύλια ήταν ταυτόχρονα και μία από τις χώρες που δημιούργησε και τις λιγότερες θέσεις απασχόλησης με αυτά τα κονδύλια. Δεν ξέρω αν είναι το πρόβλημα αυτό ίδιο της Πορτογαλίας ή είναι ένα διαρθρωτικό πρόβλημα των ε, κονδυλίων της συνοχής ή των κονδυλίων για την επαγγελματική κατάρτιση. Ίσως είναι πιο γενικό αυτό το πρόβλημα. Και τέλος, για να μην μακρηγορήσω, έχω μια τέταρτη ερώτηση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη μια πολιτική συγκέντρωση των κονδυλίων για την ε, ανακύκλωση των επιχειρήσεων ή για την ενεργειακή απόδοση ή για την ε, καλύτερη πολεοδομική και χωροταξική ρύθμιση. Γιατί αυτά είναι πολύ σημαντικά εργαλεία. Γιατί λοιπόν να μην ε, εξορθολογήσουμε και να μην συγκεντρώσουμε τα διάφορα μέσα χρηματοδότηση σε ένα ενιαίο ευρύ πρόγραμμα που θα έχει ένα πολλαπλαστικό αποτέλεσμα και θα δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας και μάλιστα θέσει εργασίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό χρειαζόμαστε, ένα τέτοιο πρόγραμμα πολεοδομικής ανασυγκρότησης των πόλων. Ευχαριστώ. Από το EFD δεν βλέπω κανέναν, οπότε τελείωσαν τώρα οι τοποθετήσεις εξ ονόματος των ομάδων, οπότε Κανονικά θα μιλήσει τώρα η κυρία Χιμπνερ, αλλά έχει κολλήσει στο μποτιλιάρισμα. Εάν έρθει, όταν έρθει, βεβαίω θα λάβει τον λόγο. Έχω μακροσχελή κατάλογο συναδέλφων που ζήτησαν τον λόγο, αλλά τώρα για τον πρώτο γύρο θα ακούσουμε τον κύριο Επίτροπο έτσι ώστε σε 10 λεπτά και 8 άμα θέλετε να δώσει τις ε, πρώτες απαντήσεις και μετά θα ακολουθήσουμε τον, ε, τον κατάλογο. Και οι συνάδελφοι θα λάβουν το λόγο για δύο λεπτά. Εγώ νόμιζα ότι μου δώσατε 10 συν 8. Ήλπιζα τουλάχιστον. Εν πάση περιπτώσει. Όπω και με τον προπολογισμό. Λοιπόν, σημαντικό θέμα το οποίο έδειξε ο Γιάνν Όλμπριχτ. Η περιφερειακή πολιτική να αγγίζει όλες τις περιφέρειες, αλλιώς ε, δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την Ευρώπη 2020. γιατί έχουμε 271 περιοχές, 84 από αυτές είναι περιφέρειες συνοχής και υπολογίζουμε με βάση τα θετικά δεδομένα πως στην επόμενη περίοδο θα έχουμε 68 μόνο περιφέρειες συνοχής. Αυτό είναι βελτίωση ε, από πλευράς πληθυσμού ε, άνω των 30 εκατομμυρίων ανθρώπων με την προσθήκη αυτών των 68. Οπότε θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη κατάσταση όσον αφορά την ευημερία από ό,τι στο παρελθόν. Η αποτελεσματικότητα της πολιτικής. Αυτό είναι το αποφασιστικό. Ήδη σήμερα, και αυτό είναι απόλυτο σωστό, ήταν λάθος να παρουσιάσουμε την Ευρώπη 2020 πως ε, εάν έχουμε τελειώσει με το οικονομικό πλαίσιο έχουν τελειώσει όλα και συνέπεια θα έχει αυτό ότι το 2015-2016 ε, θα θα έχουμε καταφέρει. Όχι, δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Πρέπει να ξεκινήσουμε ήδη από τώρα να α, ε, βλέπουμε τους στόχους και σήμερα μπορούμε να πούμε πως ε, από ένα προπολογισμό 300 ε, δισεκατομμυρίων έχουμε δώσει ήδη 300 εκατομμύρια για τους στόχους της Ευρώπης 2020. Και αυτό το οποίο είναι αποφασιστικό και ε, θα πρέπει να είναι η εξέλιξη για το μέλλον είναι να δώσουμε έμφαση στην διάθεση των κονδυλίων για να έχουμε ορατότητα, αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων σε διάφορα έργα. το ευρωβαρόμετρο, έχουμε μια διπλή ευρωπαϊκή εικόνα. Έχουμε κάποιες χώρες όπου ε, υπάρχουν περιοχές συνοχής που λαμβάνουν πάρα πολλά λεφτά από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Εκεί πέρα γνωρίζει ο πληθυσμός ε, πώς χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχουμε τις άλλες χώρες από την άλλη που είναι ανταγωνιστικές ε, περιφέρειες όπου δεν είναι τόσο όρατα τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Οπότε, Κοινοβούλιο, Κομισιόν και όλοι όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να αυξήσουν την ορατότητα το, της χρήσης των ε, κονδυλίων αυτών. Οπότε ποιο είναι το θέμα να γίνουν διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη, με τις περιφέρειες, έτσι ώστε από κοινού με τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν ποιες προτεραιότητες επιλέγουν από την Ευρώπη 2020, δηλαδή, ξέρω εγώ, αύξηση των ανανεώσιμων πηγών, αλλά να πούνε από τη μία χώρες περιφέρειες και κομισιόν από την άλλη, ποια είναι η αφετηρία στην κάθε περιφέρεια, πού βρισκόμαστε δηλαδή στον τομέα αυτών και πού θέλουμε στο τέλος μιας δεκαετούς περίοδου να βρισκόμαστε στο πλαίσιο φιλόδοξων αλλά ρεαλιστικών στόχων. Αυτό πρέπει να είναι κάτι το διάφανο και άρα νομίζω πως έτσι θα αυξηθεί η πίεση για να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα. Πολλές φορές αναφέρθηκε το πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε άλλους ε, τομείς πολιτικής. Παραδείγματο χάρη είχαμε τις συζητήσεις ε, σε παλαιότερες ε, συνεδριάσεις της Επιτροπής μας. Εν το μεταξύ, εντός της νομίζω πως υπάρχει μεγάλη διάθεση οι διάφοροι τομείς πολιτικής να συνδεθούν με την περιφερειακή πολιτική και άρα ήδη είχαμε απευθύνει πριν από λίγες εβδομάδες μια πρόσκληση σε άλλες γενικές διευθύνσεις. Συνολικά έχουμε τρεις ομάδες εργασίας που κοιτάνε τους διαφορούς θεματικούς τομείς όπου λαμβάνουν χώρα διαφορές ε, συζητήσεις, δηλαδή Έχουμε μία για τον τομέα περιβάλλον ενέργεια, μία για τον τομέα έρευνα και μία τρίτη για το όλο θέμα της κινητικότητας. Αυτές είναι οι ομάδες εργασίας όπου θεματικά κάνουμε τις διαπραγματεύσεις. Τώρα πολύ επίπεδη διακυβέρνηση θα καταθέσουμε μία πρόταση που υπήρχε ήδη στους ε, κανονισμούς για το πώς ε, θα μπορέσουμε να εμπλέξουμε τοπικούς ε, και περιφερειακούς ενδιαφερόμενους. Ελπίζω λοιπόν πως μετά να έχουμε και τη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών. Να, πρέπει να έχουμε δηλαδή μια ξεκάθαρη δήλωση πως χρειαζόμαστε την βοήθεια πολλών για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε μια αποτελεσματική εφαρμογή. Προτείναμε η Επίτροπη Τσόλος, Δαμανάκη, Άντορ και εγώ ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο που θα έχουμε τους διάφορους τομείς πολιτικής ε, που θα χρηματοδοτηθούν με κονδύλια διαρθρωτικά, να α, ε, τους ενώσουμε για να έχουμε μια καλύτερη θεματική ε, σύνοχη, κάτι το οποίο είναι σημαντικό, ιδιαίτερα όσον αφορά το Ταμείο της ε, Ανάπτυξης Υπέθρου. Με ρώτησαν επίσης για την, τομή, την δομή με των περιφερειών. Ξέρετε, εμείς έχουμε προτείνει τις λεγόμενες μεταβατικές ε, περιφέρειες, γιατί έχουμε αυτές που είναι μέχρι το 75% του ΑΕΠ, μετά υπάρχουν αυτές του φυσικά της οδιακής κατάργησης και μετά υπάρχουν οι ανταγωνιστικές. Υπάρχει όμως κάποιες περιφέρειες που είναι μεταξύ 75% και 95% του κοινοτικού ΑΕΠ ε, που δεν ήταν ποτέ κάτω από το 75% αλλά θεωρούνται ανταγωνιστικές αλλά έχουν κατ' ουσίαν ε, την ε, ίδια επίδοση με κάποιες της κατηγορίας της σταδιακής κατάργησης. Και οι δύο κατηγορίες και της σταδιακής κατάργησης και αυτές που είναι μεταξύ 75 και 90% συμπεριλαμβάνουν γύρω στα 30 εκατομμύρια Ευρωπαίους και θεωρούμε πως είναι δίκαιο, ίσως όχι φτηνό, αλλά δίκαιο και ισορροπημένο και ε, οι δύο αυτές ε, περιοχές να έχουν ε, ίση μεταχείριση με στόχο να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Λογικά με λιγότερα λεφτά από ότι μια περιοχή σύγκλησης αλλά με περισσότερα από μια περιοχή ανταγωνιστική. Και βεβαίως θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει συντονισμός ε, του Ταμείου Συνοχής, του Κοινωνικού Ταμείου επιτόπου σε όλα αυτά τα Ταμεία Συνοχής, ειδικά το ταμείο με το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, έτσι ώστε να είναι στην αυτόνομη απόφαση των ε, περιφερειών να δώσουν αυτόν τον επιπρόσθετο προϋπολογισμό στις ανάγκες που εκείνες θεωρούν σημαντικότερες υπό την σκέπη της Ευρώπης 2020. Θεωρώ πως υπάρχει εκεί πέρα μία πτυχή απλοποίησης στο βαθμό που γίνεται να έχουμε δηλαδή κοινούς κανόνες και μόνο για κάποιους ε, συγκεκριμένους ε, τομείς ε, να έχουμε επιπρόσθετους ειδικού κανόνες. Επίσης, να βλέπουμε και τις ανάγκες των τελικών δικαιούχων, των τελικών χριστών δηλαδή που θα πρέπει να έχουν μία στο το δυνατόν πιο απλή πρόσβαση. Ήδη σήμερα έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό earmarking ε, που λειτουργεί γεγονός είναι πως ήταν υποχρεωτικό για τα παλαιά κράτη-μέλη και προαιρετικό για τα νέα, αλλά βλέπουμε πως και εκεί πέρα που είναι εθελοντικό τηρείται αυτή η υποχρέωση. Σημαντικό είναι το θέμα της καινοτομίας. Η καινοτομία είναι γεωγραφικός όρος, όταν μιλάμε, ενώ η έρευνα και η ανάπτυξη πάει στον τομέα της αριστείας. Οπότε πρέπει να βρούμε την σωστή μετάβαση. Υπάρχουν πάρα πολλά, υπάρχουν αρκετά λεφτά, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε προβλήματα εδώ πέρα. Θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να επανέλθω σε κάποιες ε, ερωτήσεις και ζητώ συγγνώμη να μην ε, ζητώ συγγνώμη αν δεν απάντησα σε κάποιες ερωτήσεις. Κάτι τελευταίο το οποίο αναφέρθηκε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε πώς οι περιφέρειες ε, και οι χώρες θα χρησιμοποιήσουν τα λεφτά. Να δώσω ένα παράδειγμα, την Ελλάδα. Εδώ πέρα η, τα κονδύλια της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής ε, και ε, Τράπεζας Επενδύσεων συνδέθηκε με το ότι θα πρέπει να υπάρχει συγχρηματοδότηση με το Διαρθρωτικό Ταμείο για να διασφαλίσουμε πώς τα λεφτά αυτά πράγματι θα πάνε προς την ανάπτυξη, την επένδυση στη χώρα αυτή και πράγματι το 2010 η Ελλάδα υπ' αυτή την πίεση για πρώτη φορά μπόρεσε να εξαντλήσει την προβλεπόμενη ε, ποσόστοση και με σημαντική αύξηση βεβαίως ε, των κονδυλίων που απορροφήθηκαν με τεχνική αρρωχή κτλ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Πράγματι, ναι, θα έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε άλλη μια φορά γιατί και όλοι οι υπόλοιποι που ζήτησαν το λόγο θέλουν βεβαίως να λάβουν μια απάντηση από εσάς τώρα όμως. Θα δώσουμε το λόγο στην Τανούτα Χίμπνερ, την πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, κατάφερε να ξεκολλήσει από το μποτιλιάρισμα και έχει τώρα τέσσερα λεπτά. Ε, όχι παραπάνω σας παρακαλώ, γιατί έχουμε μεγάλο κατάλογο, τον οποίο θα διαβάσω, ομιλητών, που ζήτησαν το λόγο και έχουν 1,5 λεπτό ο καθένας για να μπορέσουμε να δούμε το χρόνο. Paulsen, Derek Warren, Jürgen Klute, Lach Liberatsky, Jöran Färm, Elisabeth Schröter, Karl Hacklund, José Fernández und Elisa Ferreira. Okay. Ähm, ähm, ja, da, da, da, da, da, da. Okay, jetzt aber Danuta, bitte. Thank you. thank you very much. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι το τελευταίο χρόνο μιλήσαμε τόσο εκτενώς για τη μεταρρύθμιση πολιτικής που εγώ θα επικεντρωθώ στην ανάγκη μια σωστά πλαισιωμένης περιφερειακής πολιτικής ε, στον κοινοτικό προϋπολογισμό στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Στην Ευρώπη συμφωνούμε όλοι ότι χρειαζόμαστε μεν οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη που θα στηρίζεται όμως ε, στην ανασυγκρότηση και δεν θα γεμίζει απλώς τα κενά του ΑΕΠ που χάσαμε στα πλαίσια της κρίσης αλλά θα μας ε, φέρνει πιο κοντά στην παραγωγικότητα, σε ενισχυμένη παραγωγικότητα και σε ενισχυμένη, ανταγωνιστικότητα. Γι' αυτό θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τον κοινοτικό Προπολογισμό, τι επενδυτικέ πολιτικές που θα μα επαναπροσανατολίσουν στου στόχου, της επενδύσεις και θα υποστηρίξουν όλε τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει που χρειαζόμαστε διακαώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η πολιτική συνοχή σε αυτό ακριβώ στηρίζεται σε ό,τι αφορά τη διαχείρισή τη και τον τρόπο που έχει προγραμματιστεί αλλά και τον τρόπο που εφαρμόζεται. Και αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η αιρεσιμότητα που πρότεινε θεσπίζει κάποιους παράγοντες που δημιουργούν προϋποθέσεις για αποτελεσματικές ε, και επιτυχείς αποδοτικές πολιτικές και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία και στον κοινοτικό προπολογισμό να εφαρμόσουμε μια τέτοια επενδυτική πολιτική. Ο κοινοτικό προπολογισμό δεν είναι η οριστική λύση σε οτιδήποτε. Είναι τόσο πενιχρός που θα πρέπει να ερμηνεύεται, να προγραμματίζεται και να εφαρμόζεται με τρόπο που να λαμβάνεται υπόψη ο καταλυτικός του, να ενεργεί ο καταλυτής και να ενεργεί ταυτόχρονα και ως κινητήριος μοχλός και άρα να ενισχύει πολιτικές ε, που θα φέρνει τις επιχειρήσεις, ε, που θα αποτρέπει τις επιχειρήσεις από την ε, μετεγκατάσταση, θα έχει, επαναλαμβάνω, και καταλητικό χαρακτήρα, αλλά και χαρακτήρα κινητήριου μοχλού αυτό, αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να στηρίξουμε, τις επενδυτικές πολιτικές. Επίσης θέλουμε καλύτερο συντονισμό των εθνικών προϋπολογισμών με το κοινοτικό πρόγραμμα επενδύσεων. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε πολιτικές με παρόμοια δυνατότητα και ικανότητα. Και οι πολιτικές αυτές για τις οποίες είναι αρμόδιος ο Επίτροπος Χάν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Όχι μόνο την ερεσιμότητα, αλλά και τη συνεισφορά στις εθνικές στρατηγικές και στη στρατηγική του 2020. Αλλά και η αρχή της χρηματοδότησης μας δίνει την ευκαιρία να συντονιστούμε καλύτερα με τις εθνικές μας προτεραιότητες και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα συνέργειες. Σε ό,τι αφορά την συμπερίληψη, την έννοια αυτή της ένταξης, η σύγχρονη έννοια της συμπερίληψης δεν είναι μόνο ότι όλοι θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν τους καρπούς της κοινοτικής ολοκλήρωσης, αλλά να συμβάλλουν και όλοι στους στόχους και να ε, επομίζονται όλη την ευθύνη για τη δημιουργία ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης. Θέλουμε μια πολιτική που θα εμπλέκει όλους τους ενδιαφερόμενους και δεν θα έχει κενά ε, ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης και ελπίζουμε ότι αυτή την άποψη θα βελτιώσει τα πράγματα η πολιτική συνοχή. Όταν μιλούμε με τους επαγγελματίες, ε, μας ζητούν επενδύσεις που θα προσανατολίζονται στο, την υλοποίηση των στόχων. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε και μια κρίσιμη μάζα χρηματοδότησης. Αν ο στόχος μας είναι η οικονομική μεγέθυνση και η ανάπτυξη, θα πρέπει να θεσπίσουμε αρχές που θα εξασφαλίζουν αυτή την ελάχιστη χρηματοδότηση για να είναι αποδοτικές οι επενδύσεις, εφικτές και αποδοτικές ταυτόχρονα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στους συναδέλφους που ζήτησαν τον λόγο. Γιώργος Σταυρακάκης. Ένα μέχρι ενάμιση λεπτό το πολύ λεπούμε, αλλιώς δεν θα έχουμε μετά χρόνο να ακούσουμε τις απαντήσεις του Επιτροπού. Μέχρι εάν φτάσουμε στο ότι κάποιοι συνάδελφοι δεν θα μπορέσουν να λάβουν το λόγο, Αν θέλουν μπορούν να καταθέσουν την ερώτηση γραπτός και θα την αποστείλουμε. Όλοι οι επίτροποι πάντα λένε πως μπορούν να απαντήσουν τις ερωτήσεις και γραπτός. Λοιπόν, ξεκινήστε. Αξιότιμε κύριε Επίτροπε, όλοι συμφωνούμε ότι η πολιτική συνοχή έχει αποδεδειγμένα συμβάλει στην συνολική ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω τη ενίσχυση των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία. Ειδικότερα για την περίοδο κρίση που διανύουμε τώρα, η πολιτική συνοχή διασφαλίζει επενδυτικού πόρου, οι οποίοι με τη δημοσιονομική στενότητα δεν μπορεί να είναι μόνο εθνική. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, κύριε Πίτροπε, να σα ευχαριστήσω για τι προσωπικέ προσπάθειε που κάνατε προκειμένου να στηρίξετε τι ελληνικέ περιφέρειε να αυξήσουν το ρυθμό απορρόφηση των πόρων. Θα ήθελα να σταθώ στι προτάσει τη Επιτροπή και πρώτον στο θέμα η εξάρτηση της αποταμίευσης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων από την τήρηση μακροοικονομικών προϋποθέσεων, macroeconomic conditionality. Κύριε Επίτροπε, κατά πόσο έχει εξετάσει η Επιτροπή την πρακτική εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος, καθώς και τις συνέπειες του για τις περιφέρειες που πλήττονται στην κρίση. Και δεύτερον, όσον αφορά το θέμα αποθεματικού επίδοσης, performance reserve, και ειδικότερα στα κριτήρια με τα οποία θα γίνεται η βράβευση των περιφερειών η εφαρμογή, η εφαρμογή τους προϋποθέτει ότι θα καθορίζονται μετρήσιμοι ποσοτικοποιημένοι στόχοι στη βάση ειδικά σχεδιασμένων δικτών, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο στην πράξη. Κύριε Επίτροπε, πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να απαντήσει σε αυτές τις δυσκολίες προκειμένου να εφαρμόσει τις προτινόμενες αλλαγές. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Τέλεια. παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι μια Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει και μια εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά. Για να λειτουργεί όμως πραγματικά εύρυθμα και αποτελεσματικά αυτή η εσωτερική αγορά θα πρέπει να δώσουμε έφαση στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία γιατί το σύνολο της ευρωπαϊκής δράσης ε, στηρίζεται σε αυτή την αρχή. Είναι λοιπόν ουσιώδες όλες οι ευρωπαϊκές περιφέρειες ε, να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την πολιτική, να εμπλέκονται σε αυτήν. Βέβαια θα μπορούσε ίσως να γίνει μια διαφορετική κατανομή του ποσοστού συγχρηματοδότηση και ορισμένες περιφέρειες ε, να συμμετέχουν σε υψηλότερο βαθμό και άλλες σε λιγότερο. Αλλά σίγουρα όλες οι περιφέρειες θα πρέπει να συμμετέχουν, να μην αποκλείεται καμία. Νομίζω ότι ήμουν αρκετά λακωνική. Ευχαριστώ κύριος Ντέρεκ Γουόν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη μάχη που έδωσε για την περιφερειακή πολιτική και ελπίζω να συνεχίσει ε, απερίσπαστα τις προσπάθειές του στο μέλλον, γιατί μερικές χώρες προσβλέπουν στην πολιτική συνοχής και εμείς ε, αναφερθήκαμε ότι μετά το 2020 είχαμε επανεθνικοποίηση των διαρθρωτικών κονδυλίων. Δεν συμφωνώ με, αυτό το συμπέρασμα της πέμπτης έκθεσης συνεχής νομίζω ότι δεν θα βοηθήσουμε έτσι την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Πάντω, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σα υποστηρίξει τον αγώνα που δίνετε για την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχή. Οι περισσότεροι συνάδελφοι συμφωνούν με του γενικού προσανατολισμού τη πέμπτη έκθεση συνοχή, αλλά θα πρέπει να ρυθμίσουμε κάποιε λεπτομέρειε. Έχω μία πληθώρα ερωτημάτων, αλλά θα περιοριστώ σε δύο μόνο σήμερα το πρωί. Η πρώτη ερώτηση αφορά το θέμα των κινήτρων αποδοτικότητας ή επιδόσεων δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο να αφαιρεθούν κάποια κονδύλια από πιο αδύναμε περιοχέ και να μεταφερθούν σε κάποιες που είναι πιο ισχυρέ και έχουν περισσότερε ικανότητε. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο σωστό τρόπο. Μήπω θα μπορούσαμε να βρούμε άλλο τρόπο να δώσουμε κίνητρα, ενάυσματα στι περιφέρειε για να υλοποιήσουν ε, του στόχου του 2020 πέραν των πρημοδοτήσεων που προτείνεται. Σε ό,τι αφορά τι ε, αστικέ Είπατε ότι δεν υπάρχει ορισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τι εστί αστική περιφέρεια, αστική ζώνη. Ε, επαφίεται στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών ορισμός αυτός. Έχω όμως εδώ κάποια ανησυχία. Αν τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα. Μια στιγμή. Αν τα κράτη-μέλη ε, θεσπίσουν τον ορισμό, ίσως περιοριστούν μόνο σε μεγάλες πόλεις. Θα προτιμούσα ο ορισμός ε, να προσδιορίζεται από τις περιφέρειες και όχι από τα κράτη-μέλη. Κλούτε. Ναι, ευχαριστώ Γιούτα. Ελπίζω να είμαι σύντομος. Να τονίσω πως κατά την άποψή μας το Ταμείο Συνοχής είναι το μεγάλο κοινωνικό μέσο της Ένωσης για τη σταθεροποίηση και τη συνοχή. Επίσης να τονίσω αυτό το οποίο είπε συνάδελφος πως πρέπει να γίνει απλούστερη πρόσβαση για τους χρήστες χωρίς να υποφέρει ο έλεγχος. Το θύμα αιρεσιμότητας ε, και του αποθεματικού σύμφωνα με τις επιδόσεις το ανέφεραν ε, και προλαλήσαντες και δεν θέλω να το επαναλάβω. Πρέπει να το υπογραμμίσουμε όμως είναι σημαντικό αυτό ο στόχος του Ταμείου Συνοχής. Επίσης ακούστηκε κάτι για τρέχοντα εναλλασσόμενα ταμεία, τι είναι αυτό το πράγμα, πώς θα χρηματοδοθεί και πόσο κοστίζει και μετά για την απέτηση της ευρυζωνικότητας. Δεν ξέρω εάν θα πρέπει ε, να προωθήσουμε κάτι τέτοιο στις περισσότερες χώρες Ένωσης. Ε, εν τω μεταξύ, καλά πάντα πράγματα και από πλευρά εξοπλισμού, η βιομηχανία, ο κλάδος επενδύει. Είναι κλάδος κλάδο, ε, δεν ξέρω, στον οποίο εάν πρέπει να ενισχύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Μπόγκουσλαβ Λιμπεράτσκι τώρα. Eh, Κύριε Επίτροπε, γεγονό, γενικά ε, είμαι ικανοποιημένο με αυτά που άκουσα από εσά και συμφωνώ με αυτά που είπε και η κυρία Κωνσταντζα Κρέλ. Εγώ θα ήθελα να ενισχυθούν οι κοινωτικέ μέθοδοι σε ό,τι αφορά την βελτίωση των προβλημάτων και θα πρέπει να στηριχθούμε στην ε, συνοχή και την αλληλεγγύη που είναι ακρογωνία η λύθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα των υποδομών. Τι μοντέλο πιστεύετε ότι είναι το ιδανικό. Πιστεύουμε ότι τα χρήματα θα πρέπει να αξιοποιούνται σωστά, να πιάνουν τόπο. Και με διαφανή και ορατό τρόπο να αξιοποιούνται και μάλιστα να ικανοποιούν τι προσδοκίε των, ε, των Ευρωπαίων πολιτών. Έχουμε 10 δισεκατομμύρια για τι υποδομέ. Έχουμε όμως 10, έχουμε 10 ε, δισεκατομμύρια που θα χρησιμοποιηθούν ε, για τις αυτοκινητοδρόμους και με τι ε, μοντέλο, με τι, ποιο μοντέλο πιστεύετε θα δώσει την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση αυτών των κονδυλίων σε ό,τι αφορά τη δημιουργία αυτοκινητοδρόμου για παράδειγμα. Επίσης θα πρέπει να εφαρμόσουμε την ε, πρακτική αρχή use or lose, δηλαδή αν κάποιος δεν είναι στη θέση να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια να τα χάνει. Νομίζω ότι καλό είναι τα κονδύλια να αξιοποιούνται από τις περιφέρειες που έχουν την ικανότητα να τα χρησιμοποιούν. Νομίζω τελείωσε και νωρίτερα το χρόνο μου. Ευχαριστώ, Δεν θα μιλήσω ως συντονιστής αλλά σου Σουηδός. Εμείς έχουμε περαιτέρω κονδύλια λόγω το ότι έχουμε σχεδόν απεριμωμένες περιοχές και υπάρχει ένα μπόνους για αυτές τις περιοχές. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με, το, με την κατάσταση αυτών των περιοχών. Δεν είναι πολύ φτωχέ, αλλά έχουν ιδιαίτερες δημογραφικές και κλιματικές ε, προκλήσεις. Ο νέος κόσμος φεύγει λόγω του ότι δεν υπάρχουν δουλειές και εκπαίδευση. Αυτό νομίζω ότι στο πέμπτο πρόγραμμα συνοχής, στην πέμπτη έκθεση συνοχής δεν συμπεριλαμβάνεται. Ε, ποιες είναι οι προθέσεις σας ε, για αυτό το σημείο. Δεύτερον, δεν είμαι πεπισμένος από τα νούμερα που μας δείξατε για την εφαρμογή. Βλέπουμε ότι όταν προχωρούν αυτά τα προγράμματα. Έχουμε πρόβλημα με τα ανώτατα όρια ε, του δημοσιονομικού πλαισίου, ειδικά για τις πληρωμές. Και έχουμε και τρέχουσες εκρεμείς υποχρεώσεις ε, που φτάνουν στο ύψος ενός ε, ετήσιου προϋπολογισμού. Τα κράτη-μέλη αρνούνται να δεχθούν την αναγκαία αύξηση του προϋπολογισμού, αλλά αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στις πληρωμές. Δεύτερον, για την συγχρηματοδότηση. Ακόμη και αν όπως λέτε λύσατε το πρόβλημα για την Ελλάδα. Αυτή ήταν μια επιμέρους λύση και προσωρινή λύση. Μακροπρόθεσμα θα πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα. Λέτε ότι θα πρέπει να έχουμε ε, πολυάριθμους κανόνες για τη συγχρηματοδότηση. Τι ακριβώς εννοείτε, διαφοροποιημένους κανόνες. Σρέντερ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να τονίσω πως περιφερειακή πολιτική και πολιτική συνοχής και αυτή είναι η πολιτική η οποία εκμεταλλεύεται πλήρω τις συνέργειες μέσω μιας κεντρικής προσέγγισης, δηλαδή της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξία για τα κονδύλια χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό μάλιστα η Επιτροπή μας σχεδόν ομόφωνα και με την άποψη του ECR είπε πως υπάρχει μια κοινή ε, γραμμή σχεδόν με τα ίδια νούμερα τα οποία προτείνει η Κομισιόν. Στόχος δικός μας, της Επιτροπής μας, είναι ακριβώς να βελτιώσουμε αυτές τις συνέργειες, αλλά όχι να τα αφαιρέσουμε από την πολιτική συγκοινωνιών και ενέργεια. Και ε, έχει τελειώσει, θέλω να μάθω αυτή η πολιτική στην Κομισιόν για τα ε, έξτρα κονδύλια και να δούμε τι θα γίνει για την χρήση την καλύτερη των κονδυλίων και τις καλύτερες συνέργειες. Και εδώ πέρα αυτή η συνθήκη νομίζω τα αναφέρει. Δηλαδή το performance reserve είναι ο τρόπος που έχει η Κομισιόν για να εφαρμόσει αυτούς τους στόχους ε, επιτέλους. Νομίζω και η προηγούμενη επίτροπος το είχε περάσει. Δεν θα πρέπει το Κοινοβούλιο εδώ πέρα να σταθεί στο πλευρό των κρατών μελών, αλλά της Κομισιόν για να επιτύχουμε όσο δυνατόν περισσότερα. Αυτό είναι μια εσωτερική αιρεσιμότητα. Ανέφερε τις τρεις όρους αυτούς ο κύριος Επίτροπος και η μακροοικονομική αιρεσιμότητα χρησιμοποιείται λάθος. Ευχαριστώ, Καρλ Άκλουντ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι. Ε, σχολίασαν τις διάφορες θετικές στοιχές πολιτικής συνοχής. Εγώ θέλω να αφαιρθώ σε ένα πιο δυσάρεστο θέμα. Είδα κάποια έγγραφα ε, επιτάπητος στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού οι παράτυπες δαπάνες, ε, κάτι το οποίο συμβαίνει εδώ και 10 χρόνια, αλλά εξακολουθεί να απασχολεί κάποια κράτη-μέλη που έχουν προβλήματα σε αρκετά τέτοια ταμεία. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Επίτροπο τι θα κάνει στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για να αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα και να μειωθούν αυτού του είδους δαπάνε. Και ταυτόχρονα θέλω να σχολιάσετε το ότι όταν κοιτάμε την ε, ανταγωνιστικότητα, τα προβλήματα ανταγωνιστικότητα που έχουμε σε κάποια κράτη-μέλη, ως ε, κομμάτι της οικονομικής κρίσης. Αυτές είναι οι ίδιες χώρες ε, που έχουν λάβει τεράστια ποσά εδώ και δεκαετίες από τα μία συνοχής και ακόμα δεν είναι ανταγωνιστικές. Ποιος είναι ο λόγος γι' αυτό. Αυτό είναι μια γενική ερώτηση, αλλά δύσκολη. Ευχαριστώ, Κάρλα. Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρεις ε, πολύ σύντομες ερωτήσεις. ποια είναι η σχέση μεταξύ της στρατηγικής Ευρώπη 2020 με την πολιτική συνοχής. Λέμε ότι η πολιτική συνοχής είναι το συμπλήρωμα της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020. Μήπως όμως είναι αλλοσυγκρουόμενες αυτές οι δύο πολιτικές. Μήπως κινδυνεύουν να γίνουν αλλοσυγκρουόμενες. Δεν θα ήταν καλό να μιλήσουμε για τα ποσά χρηματοδότησης. Τι ποσό χρηματοδοτεί τη μία και την άλλη. Κύριε Επίτροπε, θέλετε να προωθήσετε το Ταμείο Συνοχής ε, για την πολιτική μεταφορών ε, ή ποιο άλλο ταμείο αν όχι αυτό. Ελίζα Φερέιρα. Για ένα μισή λεπτό. Δύο ερωτήσεις προς τον Επίτροπο. Ένα, για τους πολιτικούς στόχους της πολιτικής συνοχής. Μιλάτε για μεταβατικές περιφέρειες ή περιφέρειες σε μετάβαση. Και υποτίθεται ότι καλύπτονται όλες οι περιφέρειες. Μήπως θα έπρεπε τώρα να εξετάσουμε πιο προσεκτικά τις ε, περιφέρειες που έχουν διαφορετικές ε, αποκλήσεις από το μέσο κοινοτικό όρο. Είτε έχουν χρησιμοποιήσει είτε όχι τα προηγούμενα κονδύλια καλά. Μιλάμε ε, για περιφέρειες που έχουν λάβει ιδιαίτερη προσοχή, ε, για περιφέρειες που είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες κτλ. Ε, Ακόμα και τώρα, ε, περισσότερο από τώρα μάλλον, κοιτάμε τις, ε, τις αντιφάσεις των διαφόρων ε, πολιτικών. Στην δική μου περιφέρεια υπάρχουν προβλήματα υποδομών. Υπάρχει υπάρχουν επιπτώσεις αρνητικές ε, λόγω των διαφορών της φορολογικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτό πλήττεται η δική μου περιφέρεια. Καλό θα ήταν λοιπόν να θετήσουμε μια πιο προσεκτική προσέγγιση από τη μετάβαση της φάσης των υποδομών στη φάση της στρατηγικής του 2020. Γιατί για να είναι αποδοτική αυτή η στρατηγική και να ευοδοθεί θα πρέπει να εφοδιαστεί με νέα μέσα ώστε η ανάπτυξη να είναι όντω ανάπτυξη που θα γίνει με σύγκληση και όχι με σταδιακή διεύρυνση του χάσματος. Ο Λάμπερτ Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Κομισιόν για την ε, προσέγγιση της ε, για το ότι θα δει μια ενιαία προσέγγιση σε ένα πλαίσιο για τα μία θαλάσσια, ε, γεωργίες ε, κτλ. Εξαιρετικά. Ένα ε, ερώτημα έχω για τα καινοτόμα μέσα για την επένδυση. Όταν μιλάμε για επενδύσεις θα πάμε πιο πολύ προς την εγγύηση, εναλλασσόμενα ταμεία και ιδιωτική χρηματοδότηση για να πληρωθούν τα προγράμματα. Αλλά ποιος ε, θα είναι, τουλάχιστον ε, αυτό είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα πάτε κι εσείς προς την ίδια κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Γλιτώσαμε κάποια δευτερόλεπτα. Ένα λεπτοδάκι. Στις παρεμβάσεις των συναδέλφων δεν ε, ακούστηκε το θέμα των αστικών περιοχών. Το θέμα της ανάπτυξης των αστικών περιοχών έχει τεράστια επίπτωση στις περιφερειές μας. Τι πιστεύετε, Επίτροπε, για την ένταξη αστικών περιοχών ε, στα ταμεία αυτά, στο Ταμείο Συνοχής, αν προκειμένου. Ωραία, συντομότατα τώρα θα ακολουθήσει ο κύριος Επίτροπος με τις απαντήσεις. Εάν δεν απαντήσει σε κάθε ερώτηση, δεν είναι η τελευταία φορά που θα μιλήσουμε για τη μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων και τη σχετική πολιτική, οπότε ψυχραιμία. Λοιπόν, κύριε Επίτροπε, για το αποθυματικό αυτό των επιδόσεων. Ευχαριστώ για την στήριξη του Κοινοβουλίου για τις ε, σκέψεις αυτές. Ποιο είναι το θέμα. Θέλουμε να έχουμε ένα μικρό ποσό, μιλάμε για 2%, να το χρησιμοποιήσουμε για τις περιοχές εκείνες οι οποίες στο πλαίσιο των ε, συμφωνιών σε μια μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση ε, τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, καλύτερα από ό,τι είχαμε συμφωνήσει. Ε, έτσι ώστε να τις επιβραβεύσουμε οικονομικά. και δεν είναι θέμα ισχυρότερης ή ασθενέστερης ε, περιοχής, αλλά αφορά την εσωτερική εξέλιξη μιας περιφέρειας. Να δώσω ένα παράδειγμα. Εάν μια περιοχή έχει 0% ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας, ξέρετε πως ο ευρωπαϊκός στόχος είναι 20% και ο στόχος στο τέλο περίοδου είναι 10% ε, που είναι βεβαίως κάτω το μέσο όρο. Αλλά ο καθένας πρέπει να συνεισφέρει και διαπιστώνουμε στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση πως δεν έχουν φτάσει στα 10% αλλά 13%. Τότε αυτή είναι μια περιφέρεια που θεωρούμε πως ε, είναι υποψήφια για μια τέτοια διάκριση ας πούμε. Το ίδιο και για μια περιοχή που πάει από το 30, έχει στόχο ξέρω εγώ το 45 και φτάνει το 50 βλέπουμε. Έτσι ε, θέλουμε να δούμε τα πράγματα. Τώρα, αιρεσιμότητα θα πρέπει να συνδεθεί με τις ανάγκες της πολιτικής συνοχής. Το επαναλαμβάνω συνέχεια, αλλά το θέμα είναι να δούμε τα ελλείμματα τα οποία οδηγούν σε μια πιο καθερημένη εφαρμογή να παραμεριστούν. Υπάρχουν ε, χώρες που δεν έχουν ακόμα κτηματολόγιο. Ε, δεν μπορούμε να επενδύσουμε όταν δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκει η γη. Αυτό δεν είναι μόνο σημαντικό για την περιφερειακή πολιτική, αλλά για ολόκληρη την εσωτερική αγορά να γίνει κάτι τέτοιο, το να ξεπεράσουμε αυτό το, το πρόβλημα. Αστικές ζώνες. Βεβαίως από πλευράς ε, Eurostat υπάρχει ορισμός, αλλά εξαρτάται από τη δομή μιας χώρας, ε, τι θεωρεί ε, μεγάλη πόλη ή αστική περιοχή. Δηλαδή το να συγκρίνουμε τη Φιλανδία με τη Γερμανία θα δείτε πως υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες και θα πρέπει ε, άνα χώρα να κρίνουμε και να δούμε τι εννοούμε μεγάλες αστικές περιοχές. τώρα αυτό το κεφάλαιο για τα εναλλασσόμενα αυτά κεφάλαια ταμεία είναι ένα κομμάτι του προπολογισμού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί όχι υπομορφή επιδόσεων, ε, υπομορφή επιδοτήσεων αλλά υπομορφή εγγυήσεων. Υπάρχουν πολλά έργα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής όπου δημιουργείται κάποιο έσοδο. Και σωστό είναι να υπάρχουν νομίζω κάποιες πληρωμές και προς την άλλη κατεύθυνση για να ξαναχρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια για να υπάρχουν μεγαλύτερα αποτελέσματα. Για το όλο θέμα της ευρυζωνικότητας υπάρχουν ήδη περιφέρειες όπου η πρόσβαση και η διάθεση των ε, τεχνολογιών ε, ίσως ξεφεύγει από μια σκληρή απλή οικονομική ανάλυση. Βλέπετε πως υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις γιατί υπάρχουν ε, περίπλοκα επιχειρηματικά μοντέλα μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. Αν λυθούν αυτά, ε, δεν είναι πλέον το θέμα το, το πώς θα μπουν τα, τα καλώδια, αλλά είναι δύσκολη η διαδικασία. Παραδείγματο χάρη το έχω συζητήσει αυτό με πολλούς συναδελφούς και έχουμε πει πως θα πρέπει να εξαντλήσουμε εκεί πέρα τα, τα κονδύλια. Ήδη η Λιθουανία έχει επιτύχει εκπληκτικές επιδόσεις νομίζω με κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που δίνει ξέρω, σε ανάπηρους, ηλικιωμένους, σε απομακρυσμένες περιοχές πρόσβαση για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τον, τον υπολογιστή και να τους σε πάρα πολλά πράγματα. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα τώρα. Ήδη και τώρα έχουμε την δυνατότητα, δυστυχώς χρησιμοποιήθηκε λίγο πέρσι, ε, για διακοπή ε, πληρωμών. Έγινε αυτό 40 φορές ε, συνολικά και στις περισσότερες περιπτώσεις στο πλαίσιο αυτών των διακοπών μπορέσαμε να λύσουμε τα ζητήματα και δεν χρειάστηκε να φτάσουμε σε πλήρη αναστολή. Τέλος, με ρώτησαν για τα ομόλογα έργων. Αυτό είναι για μεγάλα έργα, για διεθνή ε, έργα, συγκοινωνιακά, ενεργειακά. Πρέπει να δούμε εκεί πέρα τι, πώς θα γίνει. Αλλά για την εφαρμογή θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μιλήσετε και με τους συναδέλφους Έτιγκερ και Κάλλας ε, ε, γιατί πάντα λένε πως πρέπει να το δούμε κάπως στρατηγικά γιατί μπορεί να φτιάξουμε έναν ε, ωραίο διεθνή αυτοκινητόδρομο και να μην έχει δρόμους πρόσβασης σε αυτόν. Πρέπει λοιπόν και εκεί πέρα να συνεισφέρουν και οι χώρες και οι περιφέρειες. Οπότε ε, χρειάζεται και η συνέργεια εδώ πέρα να υπενθυμίσω επίσης κάποια πράγματα για να τα αξιολογήσουμε, να τα έχετε κατά νου. Βρισκόμαστε στον τομέα της ε, περιφερειακής πολιτικής. Ε, ξέρετε πώς εξαρτώμεθα από την επικουρικότητα. Δεν είναι δυνατό να γίνονται όλα εκ Βρυξελών και να εφαρμόζονται και να επιτηρούνται. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε δύο εκατομμύρια έργα εκ Βρυξελών ορμόμενοι. Εδώ πέρα πρέπει να κινητοποιηθούν οι περιφέρειες. Τώρα το ότι κάτι λειτουργεί εδώ καλύτερα και εκεί χειρότερα, αυτό εντάξει εξαρτάται και από τα άτομα. Στόχος μας είναι συνολικά να αυξηθεί η πολιτική. Αλλά η πολιτική πρέπει να δουν τρία μεγάλα πράγματα. Πρώτα απ' όλα να μειωθούν οι αντιθέσεις που είναι ιστορικό καθήκον. Δεύτερο νεότερο το οποίο σχετίζεται κυρίως με την Ευρώπη 2020. Να επενδύσουμε με ε, βάρος περισσότερο στην ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία, μια ευρωπαϊκή ορατότητα και μια τρίτη λειτουργία που συχνά παραβλέπεται είναι αυτή η οποία προκαλεί τους περισσότερους ε, πόνο κεφάλους είναι το ότι σε πολλές χώρες ε, και περιφέρειες να αναπτύξουμε τις ε, δυνατότητες για το πώς πληρεί κανείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές, πώς εκτελεί πολυετή περίπλοκα έργα. Εδώ πέρα συχνά έχουμε ένα ρόλο ανοιχνευτεί προπομπού, δηλαδή κοιτάμε τι γίνεται με τις δημόσιες προμηθείες, με τους διαγωνισμούς, με την εφαρμογή ε, ευρωπαϊκών διατάξεων στο περιβαλλοντικό ας πούμε και εκτιμένο. Εδώ πέρα, στην περιφερειακή πολιτική πρώτα βρίσκουμε τυχή την έλλειψη και μετά ε, προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε. Και επιμένω πως Όλα αυτά τα έργα, όλε αυτέ τι επιθυμίε, δεν είπαμε τίποτα παραδείγματο χάρη για τη διασυνοριακή συνεργασία. Όλα αυτά μπορούμε να τα εφαρμόσουμε εάν έχουμε έναν α, προπολογισμό σαν και αυτόν που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλιώ τίθεται το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των κονδυλίων και, του, και της σχέσης με το διοικητικό κόστος. Οπότε Ξέρετε πως εγώ είμαι υπέρ μιας Ευρώπης των έργων και όχι των ε, διαδικασιών και ελπίζω εκεί να καταλήξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Μια σύντομη παρέμβαση από την κυρία Σοφία Κονή η οποία θέλει να λάβει πάρα πολύ γρήγορα το λόγο. Γρήγορα όμως παρακαλώ. Ε, χρειάστηκε να μιλήσω στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, γι' αυτό ήμουν απούσα πριν από λίγο. Ένα στοιχείο θέλω να, να υπογραμμίσω. Ε, περιοριζόμαστε από τους προϋπολογισμούς μας και σε εθνικό επίπεδο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή την οικονομική συγκυρία που είναι δύσκολη, όλοι θα πρέπει να επιδείξουμε εφάνταστο πνεύμα για τα ποσά που έχει στη διάθεσή της η πολιτική συνοχής. Σχετική σε απόλυτες τιμές και θα πρέπει να υπάρξει, να, να δούμε διαφορετικούς τρόπους χρηματοδότησης. Θα πρέπει να μιλήσουμε για καινοτόμια χρηματοδότηση. Γιατί να μην έχουμε, ε, παραδείγματο χάρη δάνεια με χαμηλότοκα, ε, με διαφορετικό τόκο από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, που θα επιτρέψει να αυξήσουμε την ικανότητά μας χρηματοδότηση των προγραμμάτων, μια και πρόκειται για δάνεια. Είναι σημαντικό, πέρα από τους από τους τρόπους χρηματοδότησης ε, που είναι κλασικοί που ξέρουμε μέχρι σήμερα, θα πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους προώθησης της πολιτικής ε, συνοχής, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλα έργα. Äh, Ευχαριστώ. Είναι κρίμα το ότι έπρεπε να φύγετε στο ενδιάμεσο, αλλιώ θα είχατε ακούσει πως το συζητήσαμε αυτό ακριβώς το θέμα. Και, ε, και στην Επιτροπή οπωσδήποτε στις 28 Φεβρουαρίου θα ασχοληθούμε ε, ακόμη πιο εντατικά με πιθανές νέες πηγές χρηματοδότησης. Οπότε, τώρα. Ζωζέ Μανουέλ. Ας... Ε, α, ναι, γεια σας. Ευχαριστούμε λοιπόν κύριε Πίτροπε. Ο Σαλβαδόρ έχει τον τελευταίο λόγο, παρακαλώ. <clears throat> Eh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ έστω και από μακριά πια τον Επίτροπο για την παρουσία του και τις πληροφορίες που μας έδωσε και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη συζήτηση. Ξέρετε, για μένα τον εισηγητή ήταν πολύ σημαντική αυτή η ακρόαση για την περιφερειακή πολιτική. Γιατί η περιφερειακή πολιτική, κατά τη γνώμη μου, θα είναι το κλειδί των μελλοντικών δημοσιονομικών ε, προοπτικών εξαιτία του περιφερειακού του χαρακτήρα. Και αυτό συζητούσα πριν από λίγο με τον συνάδελφο Φερνάντες. Θα καταλήξω σε γενικά συμπεράσματα. Καταρχήν για το επίπεδο χρηματοδότησης. Νομίζω ότι η πλειοψηφία στην Επιτροπή, η πλειοψηφία των μελών, αλλά και ο Επίτροπος και εγώ πιστεύουμε ότι η χρηματοδότηση της μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής θα πρέπει να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με τις ισχύουσες δημοσιονομικές προοπτικές, δεδομένου ότι και οι στόχοι μας πολλαπλασιάζονται και οι υποχρεώσεις μας. Θα πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε ότι η πολιτική συνοχής θα καλύπτει όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Ο κύριος Φέρμ έδωσε ένα πολύ απτό παράδειγμα. Εν, μια τόσο ανεπτυγμένη χώρα όπως η Σουηδία Χρειάζεται όλα αυτά την πολιτική συνοχή, γιατί ακόμη και στη Σουηδία υπάρχουν μειονεκτούσε περιοχέ. Και αυτή είναι η περίτρανη απόδειξη τη επιτακτική ανάγκη να έχει πανευρωπαϊκό χαρακτήρα η πολιτική συνοχή και να καλύπτει το σύνολο τη ευρωπαϊκή επικράτεια. Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική του 2020, είναι σαφέ ότι η πολιτική συνοχή συμβάλλει τα μάλα στην υλοποίηση των τριών στόχων της πολιτικής 20 2020 Smart Sustainable Inclusive Growth, FEE, βιώσιμη, ε, e, ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη και ανάπτυξη που δεν θα αποκλείει κανέναν. Δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στους πρώτους δύο, στα πρώτα δύο χαρακτηριστικά, το Smart και το Sustainable, το βιώσιμο χαρακτήρα και τον ευφύ e χαρακτήρα της ανάπτυξης, αλλά να λάβουμε υπόψη και την ανάγκη να μην αποκλείεται κανένας από την ανάπτυξη αυτή και θα πρέπει να προσδώσουμε έναν οριζόντιο χαρακτήρα και στον προϋπολογισμό σε αυτό το θέμα της συμπερίληψης. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει η στρατηγική μας να προσανατολίζεται στην υλοποίηση των, στόχων της στρατηγικής του 2020 και αυτό με ένα βελτιωμένο σύστημα σε σχέση με το ισχύον σύστημα της εξειδικευσης του earmarking που εφαρμόζεται. Ο Επίτροπος μας ανέλησε αρκετά διεξοδικά το σύστημα που στηρίζεται στην θεματική, θεματολογική συγκέντρωση των ε, κονδυλίων και αυτό το πετυχάνουμε με τις ε, αναπτυξιακές συμβάσεις που θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλους τους κοινωνικούς τομείς και ε, επαγγελματίες αλλά και τη διοίκηση σε όλα τις τα επίπεδα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δεχτούν κάποια κριτήρια αιρεσιμότητας για τη χρήση ε, των κονδυλίων στο έδαφος τους. Οπότε φαίνεται ότι οδεύουμε προς μια πολιτική που προσανατολίζεται προς τα αποτελέσματα, όπως ε, μας είπε και ο Επίτροπος ε, Αρμόδιος για τη Γεωργία και στην γεωργική πολιτική ο προσανατολισμός θα δοθεί στα αποτελέσματα και νομίζω ότι αυτή είναι και η σωστή προσέγγιση για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Είναι προφανές ότι και η περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να κρατήσει τον εδαφικό της αντίκτυπο, γιατί αυτός είναι ο θεμελιώδης στόχος της περιφερειακής πολιτικής. Φυσικά χρειάζεται συντονισμός όλων των διαρθρωτικών κονδυλίων της, των κονδυλίων της συνοχής, περιφερειακής ανάπτυξης, αλίας, χάρη σε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο που θα στηρίζεται σε αυτή την πρόταση που έγινε δεκτή με ενθουσιασμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Επίτροπος τάχθηκε υπέρ φυσικά της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που θα είναι η νευραλική διαδικασία για να επισημάνει την αποτελεσματικότητα και τη συνεισφορά της ε, πολιτικής συνοχής και ο δεύτερος βασικός κανόνας είναι η κοινοτική μέθοδος, όπως είπε ο κ. Λιμπεράσκη, που για μας είναι προτεραιότητα. Η αιρεσιμότητα θα πρέπει να ε, προσδιοριστεί καλύτερα και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χρειαζόμαστε καλύτερη χρήση των κονδυλίων. Ο δημοσιονομικός έλεγχος επίσης είναι απαραίτητο στοιχείο και ο Επίτροπος μας είπε ότι έγινε, έλαβα χώρα και κάποιες διακοπές πληρωμών, αναστολές πληρωμών. Σίγουρα για να είμαστε αξιόπιστοι χρειαζόμαστε και έναν αυστηρό δημοσιονομικό έλεγχο. Και η πολιτική συνοχή και τα διαρθρωτικά κονδύλια θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία δαπανών. Ως προς τη διάρκεια συμφωνούμε για την επταετία και Είμαστε υπέρ της απλούστευσης και ανησυχούμε για τους διαφόρους ορισμούς της αστικής ζώνης και τους στόχους ως προς αυτή κάποιους ορισμούς που είναι κάπως ασαφείς μέχρι στιγμής. Σε λίγες εβδομάδες θα λάβετε και το προσχέδιο της έκθεσης ε, με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Σαλβαδόρ. Κοιτάω το ρολόι. Λοιπόν, κοίτα, το χρόνο τον οποίο ξεπέρασε θα τον πάρουμε από την ε, εισαγωγική δήλωση. Λοιπόν, χαιρετίζω με νεύματα βεβαίως και σιωπηρά το έκανα πριν τον ε, Επίτροπο, τον κύριο Λάσλο Άντορ. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Πρώτα απ' όλα μαζί σας βεβαίως θέλουμε να συζητήσουμε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και πώς εντάσσεται και πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί για τις επόμενες δημοσιονομικές ε, προοπτικές. Το θέμα, όπως ε, έχω ήδη πει, ε, θα εξελιχθεί όπως και πριν. Δηλαδή, ο εισηγητή θα έχει τον λόγο για τέσσερα λεπτά για μια αρχική δήλωση και ο Επίτροπος μετά θα έχει 10 λεπτά και μετά θα περάσουμε στους ομιλητέ ξενόματος των ομάδων και μετά μπορούν όλοι οι συνάδελφοι να λάβουν το λόγο. Εάν Ε, θέλει κάποιο να ακολουθήσει, βεβαίω θα ακολουθήσει μετά του ομιλητέ των ομάδων. Πρώτα απ' όλα όμω, για τέσσερα λεπτά τώρα θα ακούσουμε τον Σαλβαδόρ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μην εξαντλήσω καν το τετράλεπτο. Να καλωσορίσω καταρχήν τον αρμόδιο επίτροπο Άντορ και να τον ευχαριστήσω για την έλευση του στην Επιτροπή μας αμέσω μετά την ακρόση που είχαμε με τον Επίτροπο Χάν. Εξετάζουμε εδώ τη σχέση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και την ενίσχυση της απασχόλησης στις 27 χώρες μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης εξετάζουμε τη χρήση που κάνουν οι περιφέρειες, τα κράτη και η Επιτροπή των 80 δισεκατομμυρίων που προέβλεπαν ε, τα, που έβλεπε το Ταμείο καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου προγραμματισμού. Η ομαδοποίηση των ταμείων, κατά τη γνώμη μας, μπορεί να συμβάλλει στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής συνοχής. Αυτό ήταν το συμπέρασμα που έτυχε γενική αποδοχή στην προηγούμενη συζήτηση, παρουσία του Επιτρόπου Χάν. Ο συντονισμός όμως μας είπαν ότι θα γίνει μέσω αυτών των συμβάσεων αναπτυξιακής εταιρική σχέσης. Οι συμβάσεις αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζουν τον καλύτερο δυνατό συντονισμό άσχετα με την κατηγορία των δαπανών στην οποία εμπίπτουν τα κονδύλια αυτά. Στην πέμπτη έκθεση συνοχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει στην επιτακτική ανάγκη καλύτερου συντονισμού του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, γιατί αυτά τα δύο ταμεία είναι συμπληρωματικά. Δεν θα πρέπει λοιπόν να επιτρέπουμε επικαλύψει μεταξύ τους. Ερωτώ λοιπόν τον Επίτροπο. Πιστεύετε ότι για λόγους προγραμματισμού, δημοσιονομικού προγραμματισμού, είναι σκόπιμο να ομαδοποιήσουμε όλα τα διαρθρωτικά το ταμεία και τα κονδύλια του στην ίδια κατηγορία δαπανών, δηλαδή το Ταμείο συνοχή το ΦΕΝΤΕΡ, το Γεωργικό Ταμείο, το Ταμείο Αλίας, πιστεύετε ότι θα και το Κοινωνικό Ταμείο να συμπεριληφθούν στην ίδια κατηγορία δαπανών. Και ποιο κατά τη γνώμη σα είναι ο απαραίτητο ή ο ιδανικό, ε, ε, όγκο, το ύψο, δηλαδή Τη πρικοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Δυστυχώ δεν έχω ρολόι, κυρία Πρόεδρε, οπότε δεν ξέρω πόσο χρόνο μίλησα. Ευχαριστώ. Για καλή σα τύχη ξεχάσαμε να προγραμματίσουμε και το ρολόι, οπότε δεν ξέρω πόσο μιλήσετε. Ο Επίτροπο έχει το λόγο. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσουμε μαζί τις πολιτικές και δημοσιονομικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την, τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Με τη νέα δημοσιονομική περίοδο που φτάνει, έχουμε μεγαλύτερες ευκαιρίες να δείξουμε το ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να αυξήσουμε περισσότερο την προσθέμενη αξία του προπολογισμού της Ένωσης. Δεν θα είναι εύκολο σε περίοδο ε, λιτότητας, σε περίοδο σκεπτικισμού για τις δημόσιες πολιτικές και σε περίοδο αμφισβήτησης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα, αυτό, ε, παρ όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό, ακόμα πιο σημαντικό, να έχουμε μια θαραλέα πρόταση που μπορεί να δείξει ότι η Ένωση μπορεί να είναι τμήμα της λύσης ε, στα σημερινά προβλήματα. Ο διάλογος μαζί σας ε, είναι σημαντικός γιατί εσείς απεικονείτε τις απόψεις των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι σημαντικό αυτό αν θέλουμε να υλοποιήσουμε τις προσδοκίες τους. Είμαι πεπισμένο ότι το τμήμα του κοινοτικού προπολογισμού που βοηθάει να απεμπλακεί το κλειδωμένο δυναμικό των ε, περιοχών του λαού ε, θα μας βοηθήσει να προωθήσουμε και την αλληλεγγύη φτωχών και πλουσίων και νομίζω ότι θα πρέπει να έχει και τη γενική υποστήριξη. Ε, η πρόσφατη έκθεση συνοχής και αξιολογήσεις που κάναμε δείχνουν ξεκάθαρα το θετικό ρόλο που μπορεί να παίξει η πολιτική συνοχής και το έχει ήδη κάνει προς όφελος όλων των περιφερειών και εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Η πολιτική συνοχή θα πρέπει να συνεχίσει να έχει το δικό της προπολογισμό που ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες, τις πολιτικές και τις οικονομικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Όμω θα πρέπει να βελτιώσουμε το σχεδιασμό της πολιτικής για να εξυπηρετήσουμε πιο αποτελεσματικά αυτό το στόχο. Με το Johannes Χάν ε, συζητήσατε την προσαρμογή αυτή και δεν θα επαναλάβω αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τη σημασία που δίνω εγώ προσωπικά στην αύξηση της θετική επίπτωσης των επενδύσεων αυτών. Ο πρώτος τρόπος και ο καλύτερος είναι να ξεκαθαρίσουμε και να καταλάβουν όλοι ότι η πολιτική συνοχής δεν σημαίνει απλώς περισσότερα κονδύλια. Θα πρέπει να θεωρηθεί ως μέσο για να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Έχουμε ήδη κάνει πολλά προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Ένα πιο στενό σύνδεσμος με, τις, με τους κοινού στόχους της Ευρώπης 2020, ε, ε, μεγαλύτερη εστίαση στα βασικά θέματα, μεγαλύτερη διασύνδεση με τις ε, ρυθμιστικές κανονιστικές πολιτικές και στο θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, μεγαλύτερη εμπλοκή όλων των διαφορεμένων και φορέων στο σχεδιασμό των προγραμμάτων και μεγαλύτερος προσανατολισμός στα αποτελέσματα παρά μόνο το να μας ενδιαφέρει πώς θα ξοδέψουμε τα χρήματα. Ξέρω ότι, πολύ, ότι όλα αυτά εύκολα τα λέμε, αλλά δύσκολα τα κάνουμε. Είμαι πεπισμένος ότι έχω την υποστήριξή σας και με το βιβλίο των ιδεών σας μπορούμε να πετύχουμε αυτή την πρόοδο. Θα ήθελα τώρα να πάω πιο συγκεκριμένα στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού, ε, Κοινωνικού συγγνώμη, Ταμείου. Καταρχάς, σημερι... θέλω να σας πω ότι η πεποίθησή μου είναι για να πετύχουμε την ε, συνοχή οικονομική, κοινωνική και εδαφική. Ε, για να το κάνουμε αυτό, ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις κοινωνικές, οικονομικές κτλ. που αντιμετωπίζουμε. είναι, αυτό είναι και στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και βασίζεται σε βιώσιμη, έξυπνη και μακροχρόνια ανάπτυξη. Οι σημερινές προκλήσεις δεν είναι να προωθήσουμε τις βραχυπρόθεσμες ε, προτεραιότητες που αναφέρει η πρόσφατη επισκόπηση ε, ανάπτυξης, αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα σταθερό μακροοικονομικό πλαίσιο και να εθαρρύνουμε την ανάπτυξη. Επίσης, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μέλλον όπου μπορούμε να απεμπλέξουμε το δυναμικό που έχουν τα κράτη-μέλη, η κάθε περιοχή, ο κάθε πολίτης, ε, βοηθώντας τις κοινωνίες μας και τα δύναμα μέλη τους. Από τη δημιουργία της το 1975, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ε, βοήθησε εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες να αποκτήσουν νέα προσόντα και να βρουν ε, νέες θέσεις απασχόλησης. Επίσης, ήταν ένα συγκεκριμένο παράδειγμα του πώς ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί στην πράξη την ανάπτυξη μέσω της κοινωνικής συνοχής. Η αποστολή που ορίζεται από την συνθήκη την καθιστά βασικό εργαλείο για την ε, απασχόληση, τη μείωση της στόχιας που είναι βασικές προτεραιότητες της ε, στρατηγικής 2020. Το δυναμικό του κοινωνικού ταμείου νομίζω ότι έχει αποδειχθεί. Πρώτον, μέσω των χρημάτων που επενδύει στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική ε, Απασχόλησης, ξοδεύοντας πολύ περισσότερα αναλογικά στις στοχές χώρες και επιτρέποντάς τους έτσι να αναπτύξουν το οικονομικό του δυναμικό, την κοινωνική του συνοχή, παρά αν δεν υπήρχαν αυτά κονδύλια του κοινωνικού ταμείου. Δεύτερον, η παρουσία του κοινωνικού ταμείου, οι προτεραιότητες και οι μηχανισμοί που λειτουργεί έχουν ποιοτικό θετικό αποτέλεσμα σε όλα τα κράτη-μέλη στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη, στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα και στις ε, μεταρρυθμίσεις τους. Ε, τρίτον, το Κοινωνικό Ταμείο παίζει σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση των καινοτόμων ε, προσεγγίσεων και βελτιώνοντα ε, την συνολική διακυβέρνηση. Όπω ξέρετε, το Κοινωνικό Ταμείο έχει το δικό του καθήκον, τα δικά του, τους δικούς του στόχου. Υπάρχει λόγος που δημιουργήθηκε και αυτός ο λόγος δεν έχει εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα μάλιστα, τον επενδύσουμε στου ανθρώπινου πόρους και στην κοινωνική συνοχή ποτέ δεν ήταν πιο σημαντικό από ότι σήμερα ε, στον κόσμο το παγκοσμιοποιημένο που περνάει αυτή τη δύσκολη περίοδο μετά την κρίση. Είναι ένα εργαλείο κατεξοχήν για να υποστηρίξει την στρατηγική Ευρώπη 2020 και θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί απόλυτα με αυτή και να εστιάσει τους στόχους της αυξάνοντας το ποσοστό απασχόλησης, μειώνοντας τη φτώχεια και δυναμώνοντας τα επίπεδα εκπαίδευσης. Φυσικά μπορεί αυτό το ταμείο να υλοποιήσει καλύτερα τους στόχους του μόνο όταν ε, υπάρχει συνέργεια με όλα τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά μέσα σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο. Η Ευρώπη 2020 είναι μια πλήρη στρατηγική και αυτό που χρειαζόμαστε για να υποστηρίξουμε την υλοποίηση των στόχων είναι μια πλήρης ε, εμπεριστατωμένη πολιτική. Γι' αυτό πιστεύω ότι το Ταμείο αυτό θα πρέπει να αποτελέσει, να εξακολουθεί να αποτελεί τμήμα ε, του οπλοστασίου ε, τη πολιτική ε, συνοχή. Για να το εκμεταλλευτούμε καλύτερα θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνέργεια με όλα τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά μέσα τη Ένωση, το Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξη, το Ταμείο Συνοχή αλλά και το Ταμείο ανάπτυξη Υπέθρου, Υπαίθρου, καθώς και μερικά από τα υπόλοιπα ταμεία μα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα κανονικό καλό πλαίσιο στρατηγικής για να υπάρξει συντονισμός. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει και ένα συμβόλαιο για τις επενδύσεις ε, σε ευρία βάση. Επίσης, η συμπληρωματικότητα θα πρέπει να ενισχυθεί, διευκρινίζοντας καλύτερα το πλαίσιο και τους κανόνες επιλεξιμότητας του Ταμείου και σε σχέση με τα υπόλοιπα. Θα μειωθούν έτσι οι επικαλύψεις μεταξύ των Ταμείων και των προγραμμάτων και θα απλουστευτεί η ζωή των τελικών δικαιούχων. Είμαι πεπισμένο επίση ότι η πυκλομορφία των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες είναι τέτοια που το, ταμείο, το κοινωνικό ταμείο θα πρέπει να διατηρήσει ένα, μια ευρεία εμβέλεια για, το είδο των μέτρων που μπορεί να υποστηρίξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να υποστηρίξει τα πάντα και παντού. Αντίθετα, Όπω είπα, η συγκέντρωση στι βασικέ προκλήσει τη κάθε χώρα και τη κάθε περιφέρεια είναι εκ των κάνευ. Κυρίες και κύριοι, καταλάβατε ότι πεπισμένος ότι το κοινωνικό ταμείο μπορεί και πρέπει να παίξει ένα βασικό ρόλο την επόμενη δεκαετία για να υποστηρίξει την ε, κοινοτική στρατηγική ανάπτυξη και να τονώσει την ε, κοινωνική, οικονομική και ταφική συνοχή. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν ο προπολογισμό ε, του ταμείου αυτού είναι στο ύψος των φιλοδοξιών μας. Η Κομισιόν στην ανακοίνωση για την ε, αναθεώρηση του προπολογισμού, αυτό σημαίνει ότι τα κονδύλια του ε, Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πρέπει να είναι πιο προβλέψιμα. Αυτό απηχεί την πεποίθηση και ελπίζω να συμφωνείτε ότι αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς και αξιόπιστοι με τις πολιτικές μας προτεραιότητες, θα πρέπει να αντιστρέψουμε την αρνητική τάση που υπήρχε τα τελευταία 20 χρόνια, όπου δηλαδή το μερίδιο του Κοινωνικού Ταμείου μειώθηκε από 40% ε, στο 1990 στο 22% ε, τα 100 τη σημερινή περίοδο, στη συνολική δηλαδή πολιτική συνοχή. Εξετάζουμε τώρα διάφορες δυνατότητες που έχουμε για να το πετύχουμε. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και θα χρειαστούν περαιτέρω συζητήσεις πριν να αποφασίσει και να προτείνει ε, με τα λόγου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χωρίς να σας περιγράψω με λεπτομέρειες τα σενάρια, θέλω να σας πω ότι κάθε κρατός μέλος θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις δικές του επενδυτικές ανάγκες. Ο τρόπος που θα εξελιχθεί το κοινωνικό ταμείο θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο τρόπος που δίνουν τα κονδύλια ανταποκρίνεται στις πολιτικές προτεραιότητες και επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις σε κοινωτικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο ε, στα πλαίσια των στόχων της στρατηγικής 2020. Θέλω να ακούσω τις απόψεις σας γιατί πολύ περισσότερο εσείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παίξετε πιο σημαντικό ρόλο για να καθορίσετε τις βασικές αρχές των δημοσιονομικών προοπτικών στο μέλλον σε αφορά στα πλαίσια της διαθεσμικής συμφωνίας. Επίσης ξέρω ότι αν έχουμε ένα έτσι στεναρό ποσό, πρέπει να αποδείξουμε ότι θα το ξοδέψουμε ε, με καλό και συντονισμένο τρόπο. Θα πρέπει να συγκεντρωθούμε σε συγκεκριμένες προτεραιότητες. Αυτό όμως είναι ένας τομέας. Δεν αρκεί αυτό αν δεν έχουμε και μηχανισμούς ούτως ώστε ε, να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα επιτόπου. Από το 2007 κάναμε σημαντική πρόοδο. Οι κανόνες οι εφαρμοστικοί έχουν απλουστευτεί και επίσης και τα σφάλματα σε ό,τι αφορά τις ε, επιστροφές έχουν μειωθεί και τις πληρωμές έχουν ε, μειωθεί. Αλλά θα πρέπει να βελτιώσουμε τα ποσοστά απορρόφησης ε, σε σχέση με την ποιότητα και την ποιότητα των προγραμμάτων. Ε, συχνά, λόγω της περιπλοκότητας των κανόνων, άνθρωποι μπορούν να μας βοηθήσουν προς αυτούς τους στόχους, αποκλείονται αυτό δεν είναι αποδεκτό και θα το αλλάξουμε. Για να κλείσω αυτή την εισαγωγική μου παρουσίαση, θα ήθελα να τονίσω τις τρεις κατευθύνσεις που θα ήθελα να μας απασχολήσουν. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να κατευθυνόμαστε προς μια κατεύθυνση που εστιάζεται στο ατελικό αποτέλεσμα. Επίσης θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα χωρίς να υποσκάψουμε την ασφάλεια και την κανονικότητα των δαπανών. Τρίτον, θα πρέπει να υλοποιήσουμε περισσότερο και να ασχοληθούμε περισσότερο με την αναλογικότητα. Αυτοί είναι οι τρεις ε, άξονες που θα υποστηρίξουν τις μελλοντικέ προτάσεις της Κομισιόν. Αν κάνουμε το σωστό, μπορούμε να βγούμε από αυτή τη συζήτηση με μια πιο ισχυρή πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι δεχόμαστε και την ανάγκη όμω για προσαρμογή. Σημαίνει ότι θα κάνουμε επιλογέ. Σημαίνει ότι θα έχουμε το θάρρο να αλλάξουμε τα πράγματα τα οποία μέχρι στιγμή δεν πήγαν τόσο καλά. Είμαι πεπισμένο ότι μαζί μπορούμε να καταστήσουμε ε, ισχυρό εργαλείο την πολιτική συνοχή, ούτω ώστε η Ευρώπη να βγει μια και καλή από την κρίση και να μπει στο, στην πορεία τη έξυπνη. Ε, βιώσιμης και ε, με συμμετοχή όλων ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Αυτή ήταν η ερμηνεία της Επιτροπής για το τι σημαίνει δεκάλεπτο. Πριν περάσουμε στο γύρο των εκπροσώπων των ομάδων, θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά την, τον πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Κάποια στιγμή φυσικά θα φύγει δεν θα παρακολουθήσω όλη τη συζήτηση, αλλά θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον κύριο Λαμασούρ, τον πρόεδρο της Επιτροπής. Εκτός ότι θα ήθελα να το ευχηθώ ε, χρόνια πολλά, γιατί έχετε γενέθλιά του ο Λαμασούρ. Και τώρα μπορώ να περάσω στους εκπροσώπους των ε, ομάδων. Νομίζω ότι το καλύτερο δώρο για τα γενέθλια του κ. Λαμασούρ θα ήταν να εγκρίνουμε του ίδιου πόρου. Ω εκπρόσωπο του ΕΛΚ θα ήθελα απλώ να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό ότι έχουμε την ίδια μέρα δύο επιτρόπου να ασχολούνται με την ίδια πολιτική. Γιατί έχουμε μιλήσει επανειλημμένω για τη σημασία τη πολιτική αυτή, στο επίπεδο τη χρηματοδότηση, την αποδοτικότητα που θα πρέπει να είναι το μέλημα και των δύο επιτρόπων. Οπότε είναι σημαντική η σημερινή ακρόαση. Αναπόφευκτα φτάνουμε και στο πρόβλημα του συντονισμού. Και εδώ ανακύπτει το πολιτικό ζήτημα. Τι μορφή θα έχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, τι σημαίνει ολοκληρωμένη προσέγγιση, ολοκληρωμένη σε επίπεδο Βρυξελών ή θέλουμε καλύτερη ολοκλήρωση των δικαιούχων μεταξύ τους. Πρόκειται για διαφορετικές φιλοσοφίες. Κύριε Πίτροπε, Έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ποια είναι η γνώμη σας για, το, για τη σημερινή κατάσταση του, του ενός ταμείου. Πιστεύετε ότι το σύστημα αυτό είναι αποτελεσματικό σε εθνικό επίπεδο. Γιατί νομίζω έτσι καταλήξαμε σε ένα κατακαιρματισμό ανατομέα των διαφόρων προγραμμάτων. Ποια είναι η γνώμη σας για τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε αυτές τις συμβάσεις αναπτυξιακής εταιρικής σχέσης. Θα πρέπει να είναι και το Κοινωνικό Ταμείο τμήμα της συμβάσεως με τις ανάλογε ανάλογες συνέπειες. Και υπάρχει και το ερώτημα που συνδέεται με την παρατήρηση που κάνατε προηγουμένως πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ταμείων και με σαφή προσδιορισμό των κονδυλίων. Σε ποιο επίπεδο όμως πιστεύετε θα πρέπει να προσδιορίζονται τα κονδύλια, στο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο ή στον ετήσιο προϋπολογισμό. Γιατί αυτό θα καθορίσει και το πώς θα λυθούν υπόψη προτεραιότητες. Και φυσικά ό,τι λέμε για την ε, πολιτική συνοχή ισχύει και για τα δύο σκέλη. Ευχαριστώ, Derek Γουάν για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ήμουν ανέκαθεν ένθερμος υπέρμαχος ε, των δαπανών των κονδυλίων του Κοινωνικού Ταμείου στις υποδομές για τη δημιουργία μεγέθυνσης και θέσεων απασχόληση. Αλλά φυσικά χρειαζόμαστε εξειδικευμένους ανθρώπους ε, με προσόντα και δεξιότητες που θα κάνουν σωστά το έργο τους. Γι' αυτό και είναι σημαντικό το κοινωνικό ταμείο στην Ουαλία, αλλά και αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολλά παραδείγματα χρήσης του κοινωνικού ταμείου για να βελτιωθούν οι δεξιότητες, τα προσόντα και να αυξηθεί η συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Και σήμερα είναι ακόμη πιο σημαντικό το κοινωνικό ταμείο Δεδομένη της περικοπής των κοινωνικών δαπανών και τη ε, έξαρση τη ανεργία. Θα πρέπει τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει μια δραστήρια πολιτική υπέρ τη απασχόλησης και υπέρ τη οικονομικής μεγέθυνση στο μέλλον. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να, αποτελέσει, να παραμείνει τμήμα τη πολιτική συνοχή και χαίρομαι που το δέχεται αυτό και ο επίτροπο. Φυσικά, ε, καλό θα είναι να έχουμε αποτελεσματικότερο συντονισμό μεταξύ όλων των ταμείων, αλλά αν θέλουμε περισσότερε θέσει απασχόληση, θέλουμε και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που θα αναλαμβάνει αυτέ τι θέσει εργασία. Σε ό,τι αφορά το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, εμεί δίνουμε μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ του Κοινωνικού Ταμείου. Πολλοί δίνουν μάχη για την γεωρική πολιτική, άλλε πολιτικέ, αλλά κατά τη γνώμη μου ε, η οικονομική ανάπτυξη, η μεγέθυνση και η θέση απασχόληση θα πρέπει να είναι προτεραιότητα και να φαίνεται αυτό και σε επόμενε δημοσιονομικέ προοπτικέ. Μέχρι στιγμή ε, μιλήσαμε κυρίω για το κοινωνικό ταμείο. Υπάρχουν όμω και άλλα σχέδια και προγράμματα που είναι εξίσου σημαντικά στον τομέα τη απασχόληση, τη παιδεία, διαβίου κατάρτιση. Όλε αυτέ οι πολιτικέ συμβάλλουν στην ε, υλοποίηση των στόχων τη μεγέθυνση και τη ε, αύξηση των θέσεων εργασιών στο μέλλον. Τέλος κύριε Επίτροπε, μια ερώτηση. Φαίνεται το ίδιο επίπεδο κονδυλίων θα πρέπει να δοθεί και στο μέλλον στην πολιτική συνοχή. Να μην μειωθούν τα κονδύλια τη συνοχή στο μέλλον. Έχετε κατά νου ένα ποσοστό για τι δαπάνε Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πολιτική συνοχή και στα διαρθρωτικά ταμεία σε επόμενε δημοσιονομικέ προοπτικέ. Και ένα πιο συγκεκριμένο ερώτημα για τι περιφέρειες. Σε πολλέ περιφέρειες έχουμε πολλά προγράμματα και σχέδια για κατάρτιση, επαγγελματική επιμόρφωση και είναι παρόμοια σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα σχέδια και τα προγράμματα. Μερικές φορές όμως λαμβάνει η χώρα μια επικάλυψη. Πώς θα την περιορίσουμε στο μέλλον για να συνεχιστούν βέβαια αυτά τα σημαντικά προγράμματα και σχέδια, αλλά να ομαδοποιηθούν κάπως, είναι λιγότερα ίσως. Ευχαριστώ, Κάρλ, για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Επίτροπο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις απόψεις σας για το μέλλον και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Το συζητάμε εδώ και καιρό. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στην Επιτροπή Υπερπολογισμού πριν από λίγο καιρό. Θα την ξέρετε όπου τόνισε τις απόψεις του Κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα είναι ένα μέσο που διχάζει το Κοινοβούλιο. Κάποια μέλη της ομάδας μου είναι επικριτικά και για την ύπαρξη του Ταμείου αυτού. Οπότε θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας για το μέλλον του Ταμείου και το πώς θα πρέπει να διαρθρωθεί και την ανάγκη ε, ύπαρξης αυτού του Ταμείου. Χαίρομαι που αναφέρθηκε το θέμα της αλληλεπικάλυψης γιατί είναι κάτι το οποίο το έχει θίξει και η ομάδα μας. Όσον αφορά δε το ποσό που πηγαίνει στο κοινωνικό ταμείο, Είμαι σίγουρος πως κάθε επίτροπος θα έρθει και θα πει πως ο δικός του τομέας χρειάζεται τουλάχιστον αυτό το οποίο έχει σήμερα στον προπολογισμό και είναι φυσικό. Είναι σημαντικό όταν η Κομισιόν, ε, ένα επίτροπο ορίζει την ανάγκη για περισσότερα λεφτά στον τομέα του, να έχουμε ένα σαφέ ε, μήνυμα το πού θα πάνε τα λεφτά. Γιατί φοβάμαι το ότι περισσότερα χρήματα δεν θα τα βρούμε πάρα πολύ εύκολα. Αντιθέτω, έχουμε πάρα πολλές νέες ανάγκες και σκληρές διαπραγματεύσεις ε, για τον προπολογισμό. Οπότε πρέπει να έχουμε πολύ καλά επιχειρήματα για αυξήσεις σε οποιονδήποτε τομέα. Εάν είναι να έχει περισσότερα λεφτά στο μέλλον η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ελίζαμπετ για τους πράσινους. Ε, ναι, ευχαριστώ. Ο προλαλής σας δεν κατάλαβε πού πάει η αύξηση στον τομέα του κοινωνικού ταμείου, ίσως μπορώ να το εξηγήσω εγώ. Έχει δύο νομικές βάσεις στη συνθήκη το κοινωνικό ταμείο. Το ένα αφορά την πολιτική συνοχής και ο δεύτερος το κεφάλαιο της απασχόλησης και αυτή είναι η διαφωνία, δηλαδή το εάν θα το σπάσουμε ή όχι, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία και στις δύο επιτροπές και του Κοινοβουλίου στο ψήφισμα του φθινοπόρου είπε πως δεν έχει νόημα να πάει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υπό το κοινό πλαίσιο της ε, πολιτικής συνοχής. Αλλά αυτό είπε η ομάδα μας στα δύο ψηφίσματα υπό τους κανόνες του. Δηλαδή, ε, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που πρέπει να διατηρηθεί ακριβώς επειδή μιλάμε για πάρα πολύ μικρά έργα και οι κανόνες χρηματοδότησης πρέπει να είναι ιδιαίτερα, αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα για να επιτύχουμε ακριβώς αυτό το οποίο παρουσίασε και ο κύριος Επίτροπος. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Γι' αυτό η διατύπωση είναι ναι στο κοινό πλαίσιο αλλά υπό τους δικούς του κανόνες και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο βεβαίως στον κανονισμό αλλά μας υπόσχεται τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα χρήσης αυτών χρημάτων. Θεωρώ λοιπόν, ξέρετε ο Επίτροπος είπε πως η το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν πάει μόνο στην ε, συμπερίληψη, στη στήλη συμπερίληψης του 2020 αλλά και στους τρεις ε, κανόνες αυτούς δηλαδή να είναι και ε, να συμπεριλαμβάνει να είναι συνεκτικό και έξυπνο και αηφόρο γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε τίποτα για την 2020. Παραδείγματο χάρη, οι πράσινε δουλειέ, οι πράσινες ε, δουλειές και οι απαραίτητε δεξιότητες είναι ένα παράδειγμα για το έξυπνο και το αηφόρο και βεβαίω ε, και με τη συμμετοχή ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν ανέφερε ο Επίτροπος και αυτή είναι η ερώτησή μου, είναι η δυνατότητα της ρήτρα αυτής που μας δίνεται για αλληλεπικάλυψη των ταμείων, το ESF δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που αναφέρθηκε, να χρηματοδοτηθεί και από αλλού. Αυτό έγινε στην τελευταία περίοδο με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί έτσι γίνεται πιο απλή η αίτηση χρηματοδότηση έργων και μειών τη γραφειοκρατία. Θέλω να πω πως ε, δεν αναφέρθηκαν δύο σημαντικά σημεία, δηλαδή το λάθος που έγινε κατά τη δική μας άποψη, γιατί υποκύψαμε στα κράτη-μέλη στο ότι τα διεθνή έργα πήγανε στην ε, επιλογή των κρατών μιλών. Εδώ πέρα έχει κάνει η Κομισιόν λάθος, γιατί ακριβώς αυτή η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ε, μπορεί να συνεισφέρει στο ε, κοινωνικό κομμάτι και ακριβώς ε, γίνεται σαφής η διπλή στρατηγική του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και δεύτερον εκεί που παίζει σημαντικό ρόλο το Κοινωνικό Ταμείο και πρέπει να το διατηρήσουμε είναι πρώτα απ' όλα η αρχή της εταιρική σχέσης και το gender mainstreaming. Αυτό το λέει για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αλλά ισχύει και για τα δύο ταμεία οριζοντίως είναι κρίμα το ότι αυτό το κομμάτι στην πέμπτη έκθεση συνοχής παίζει τόσο μικρό ρόλο και πρέπει να βελτιωθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ρίτσαρντ για τους Ευρωπαίους συντηρητικού. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την Επιτροπή που λέει ότι είναι χαλεπή η οικονομική καιρή και σφιχτός ο προϋπολογισμός. Ερωτώ λοιπόν γιατί από αυτέ τι περιστάσει πιστεύετε κύριε Επίτροπε θα πρέπει να διευρεθεί ο υπολογισμό για τα δικά του προγράμματα. Αυτό που περιμέναμε να μα πει ο Επίτροπο είναι όχι γιατί ήθελε περισσότερα κονδύλια, αλλά πώ θα εξασφάλιζε καλύτερη αξιοποίηση των υφισταμένων κονδύλιων. Σίγουρα το κλειδί είναι η στρατηγική του 2020 που θα πρέπει να περιλαμβάνει και οικονομική, εδαφική και κοινωνική συνοχή. Και αποδεικνύοντας ότι αυτές οι πολιτικές όχι μόνο θα έχουν προστιθέμενη αξία για την οικονομία, αλλά θα έχουν προστιθέμενη αξία και για τους πολίτες, έτσι θα αποδείξουμε τη σπουδαιότητα και τη σημασία που έχουν οι πολιτικές αυτές για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό είναι το σημαντικό. Η εμπειρία μου όμω με έχει διδάξει ότι πολύ συχνά το πρόβλημα είναι ότι πολύ συχνά το κοινωνικό ταμείο δεν ευθυγραμμίστηκε με τις προτεραιότητες και τις πολιτικές δαπανών των εθνικών προϋπολογισμών και ως εκ τούτου τα κονδύλια δεν χρησιμοποιούνται αποδοτικά, δεν αξιοποιούνται δεόντως. Επαναλαμβάνω λοιπόν την έκκληση μου. Δεν θέλουμε περισσότερα κονδύλια, αύξηση των δαπανών, αλλά καλύτερη αξιοποίηση των κονδύλιων. Ευχαριστώ Κονίλια Ένστ για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Νομίζω πως συμφωνούμε πως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συνεισφέρει και θα συνεισφέρει σημαντικά για τη συνοχή στο μέλλον και δεν πρέπει να μειωθεί το ύψος του για να αποτελέσει κομμάτι της ε, συνοχής με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν. Αυτό το οποίο με ανισχύει είναι η συζήτηση για τη στρατηγική 2020. Αναρωτιέμαι πώς θα κολλήσει αυτό αφενός με το να έχουμε μια στρατηγική που σκοπεύει βεβαίως να ευνοήσει πράγματι κάποια συγκεκριμένα πράγματα, αλλά από την άλλη βεβαίως ε, να λάβουμε υπόψη και τις ιδιαιτερότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Με ενδιαφέρει λοιπόν ακριβώς αυτή η προβληματική του 2020 ε, να ακούσουμε λίγο περισσότερα πράγματα από τον κύριο Πίτρο και τον κύριο Άντερ. Κατόπιν σε πολλές χώρες και σε εμάς, στη Γερμανία, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ε, εξειδικευμένων εργατών τα τελευταία χρόνια, το οποίο διευρύνεται. Ακριβώς λοιπόν το θέμα των εξειδικευμένων εργαζομένων είναι αυτό το οποίο πρέπει να παίξει ένα μεγάλο ρόλο στο πλαίσιο αυτού του Ταμείου και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Οπότε, εργαζόμενοι και το σχετικό πρόβλημα πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και τρίτον, αυτό αναφέρεται στο τριεθνές Πολωνίας, Τσεχίας, Γερμανίας και τις ε, περιφέρειες εκεί πέρα για τα διασυνοριακά προγράμματα. και την απέτηση να απλοποιηθούν τα διασυνοριακά προγράμματα. Από εκπροσώπους περιοχής ε, ακούμε συνέχεια πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε κάποια συνεργασία μεταξύ των ε, τριών ε, περιφερειών. Πώς θα διευκολύνουμε λοιπόν το τι θα γίνει εδώ πέρα. Κατόπιν, η αρχή της ε, συνεργασίας, ε, έχουμε ασκήσει κριτική εδώ και τέσσερα χρόνια για την καλύτερη εφαρμογή της. Ε, πράγματι και η Κομισιόν ομολογεί πως πρέπει να ενισχυθεί αυτή η αρχή και βεβαίως θα είναι και πιο στοχευμένα τα ταμεία. Οπότε τι θέλει να κάνει η Κομισιόν εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ιδιαίτερα στον, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Και τέλος, είπαμε πάρα πολλά για την καταπολέμηση της στόχιας. Θέλω να πω μόνο το εξή. Μέσω της διεύρυνση της Ένωσης είναι σαφές πως ε, ο αριθμός των φτωχών περιοχών έχει αυξηθεί και πλέον όταν μιλάμε για καταπολέμηση στόχιας έχουμε μια τελείω νέα διάσταση. Οπότε θα πρέπει να ε, ενισχυθεί η πτυχή αυτή και θα ήθελα να γνωρίζω ποια σχέδια, ποια πολύ συγκεκριμένα σχέδια έχει η Κομισιόν ως προς αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, η Πρόεδρος. Το EFT δεν εκπροσωπείται το κόμμα, οπότε θα περάσουμε σε ένα πρώτο γύρο απαντήσεων. Ο κύριος Επίτροπος έχει 8 με 10 λεπτάκια ε, σύντομα όμως έτσι όπως κάναμε παλιά. Και για να δώσω την ευκαιρία στους συναδέλφους ε, να λάβουν το λόγο. Αν Γκένσεν, Γιώραν Φέρμ, Λαμασούρ. Ε, Μπάρμπαρα Ματέρα και Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες. Ωραία και μετά θα τελειώσει εδώ ο κατάλογος των ομιλητών. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ο κύριος Επίτροπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να μην ξεπεράσω το χρόνο. Ε, μην ξεχνάτε ότι άργησα κιόλας να κάνω την πρώτη μου παρέμβαση. Άρχισα αργότερα. Αλλά δεν νομίζω ότι επηρεάζει αυτό την ουσία της συζήτησης. Ε, τα θέματα που συζητάμε είναι πολύ σοβαρά και όλα συνδέονται με τις κοινωνικές και οικονομικές ε, επιπτώσεις της κρίσης. Ε, έχουμε 23 εκατομμύρια ανέργους, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός μάλλον αυξάνουν, για να μην πω αυξάνουν δραματικά σε κάποια κράτη-μέλη. Ε, ταυτόχρονα έχουμε πολύ φιλόδοξους στόχους και νομίζω ότι οι σημερινές και μεθεπόμενες συζητήσεις για τα δημοσιονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καθορίσουν την αξιοπιστία των προγραμμάτων μας και κυρίως της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Αν θέλουμε να πούμε ότι η Ευρώπη για το 2020 είναι μια στρατηγική σοβαρή και αξιόπιστη, θα πρέπει να οργανώσουμε τα μέσα και τα δημοσιονομικά μέσα που έχουμε αναλόγως αν έχουμε φιλόδοξους στόχους να αυξήσουμε το ποσοστό απασχόληση, πέσοντας και στο επίπεδο της προσφοράς και της ζήτησης και να καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό πιο αποτελεσματικά από πριν, νομίζω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε αυτές τις, αυτούς τους στόχους με ανάλογες αποφάσεις και στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι Μιλάω ή μίλησα μόνο για ποσά. Μίλησα ελάχιστα εξάλλου για τα ποσά. Κυρίως μίλησα για το πώς θα βελτιώσουμε τη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Από τον Ιούνιο που αρχίσαμε την, ε, τις διασκέψεις αυτές για την ε, κοινωνική συνοχή θα μπορούσα, και έχω μιλήσει μάλλον, για την ε, για το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τους ε, κοινωνικούς τα πόρους, κοινωνικούς πόρους με άλλους πόρους, ούτω ώστε να έχουμε πόρους από διεθνείς τράπεζες και ενδεχομένως και από τον ιδιωτικό τομέα, ούτω ώστε να έχουμε περισσότερους πόρους για να εφαρμόσουμε τις πολιτικές μας και να έχουμε έτσι την ε, Κάναμε έτσι λοιπόν πολλές συζητήσεις, αναλύσαμε τις δυνατότητε που έχουμε και νομίζω ότι σημειώνουμε πρόοδο. Έχουμε κάποιες εμπειρίες που μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και να βασιστούμε σε αυτές, αλλά το εύρος των προκλήσεων είναι ανευπροηγουμένο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο το μέγεθος, αλλά και τη δομή του προϋπολογισμού και των ταμείων. Έχουμε διάφορες συναλλακτικέ λύσεις. Θα πρέπει να τις εξετάσουμε όλες με ανοιχτό μυαλό και τελικά να αποφασίσουμε ποια είναι η πιο ευνοϊκή λύση ή λύσεις. Για το θέμα, παραδείγματο χάρη, του μονοταμιακού συστήματος ή όχι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι Μπορούμε να επιλέξουμε, μπορούμε να, διευκρινίσουμε, να διευρύνουμε το πεδίο της επιλεξιμότητας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, τόσο ώστε να υποστηρίζει μια ευρεία ανάπτυξη στις πολιτικές μας και να υπάρχουμε τη δυνατότητα ή έχουμε τη δυνατότητα μάλλον να διευκολύνουμε ένα πολυταμιακό σύστημα χρηματοδότησης της ε, πολιτικής ανάπτυξης και να συνδυάσουμε διάφορους πόρους. Εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να κάνουμε ένα κατακαιρματισμό ανατομέα. Η απασχόληση είναι ένα τομέας και το ξεκαθαρίζω αυτό. Όταν μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ως ξεχωριστό ταμείο, δεν νοούμε ότι θα κάνουμε μια, έτσι, ένα κατακαιρματισμό των τομέων. Ε, η εργατική το εργατικό δυναμικό συνεισφέρει σε κάθε τομέα της οικονομίας με οριζόντιο τρόπο. Το κοινωνικό ταμείο θα πρέπει να συμπεριληφθεί ε, στις προσπάθειες συντονισμού. Ε, χρειαζόμαστε τον ευρωπαϊκό συντονισμό, ούτω ώστε να καταλαβαίνουμε καλύτερα πώς επηρεάζουν οι πολιτικές, αλλά θα πρέπει να έχουμε και συντονισμό σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο δικαιούχων, οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν ποιες είναι οι πολιτικές, ποιοι στόχοι προωθούνται, από ποια πολιτική ε, και χρηματοδοτούνται από ποιο χρηματοδοτικό μέσο. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη διαφάνεια και σαφήνεια υπάρχει για τους δικαιούχους, για το καθήκον και την αποστολή του, καλού, του κάθε ταμείου, τόσο περισσότερες πιθανότητες είναι, έχουμε να αποφύγουμε τις καταχρήσεις των πόρων των ταμείων. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να υπάρχει μεγαλύτερη ενάργεια ε, σε ό,τι αφορά τα ταμεία. Ταυτόχρονα πρέπει να τονίσουμε ότι στην επόμενη περίοδο θα έχουμε και να αντιμετωπίσουμε νέες ε, προκλήσεις που συνδέονται με τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Το θέμα της ε, ενεργούς γύρανσης ε, των ε, πιο ηλικιωμένων εργαζομένων που συμμετέχουν στην αγορά εργασίας είναι μια τεράστια πρόκληση. Τώρα θα πρέπει να αποφασίσουμε μεταξύ των κρατών μελών για την αύξηση των ορίων ταξιοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι να είναι παρόντες στην αγορά εργασίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη διαδικασία διαβίου μάθησης και την απόκτηση προσόντων σε μεγαλύτερη ηλικία. Αυτό όμως σημαίνει περισσότερους πόρους. Και συνδέεται, κάτι που συνδέεται με τη στρατηγική 2020, 2020 θα πρέπει να ε, υποστηρίξουμε και τους στόχους ε, αηφορίας. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερες επενδύσεις σε, πράσινες, σε πράσινα προσόντα και δεξιότητες ε, για όλους τους τομείς, όχι για ένα ή δύο τομείς μόνο. Είναι μια οριζόντια προσέγγιση και το κοινωνικό ταμείο θα πρέπει να είναι ικανό να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει το κοινωνικό ταμείο να χρησιμεύει ακόμη περισσότερο για την κοινωνική ένταξη. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Καταπολέμησης της Στόχιας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, που αναφέρεται επίσης ε, τη χρηματική διάσταση και στις χρηματοδοτικές ανάγκες και έχουμε και συγκεκριμένα θέματα που θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε ε, τη συμπερίπτωση Φερρυπίν της μειονότητας των Ρωμά. Η κατάσταση σε ορισμένα κράτη-μέλη είναι δραματική σε ό,τι αφορά τους Ρωμά και το Κοινωνικό Ταμείο είναι το κατάλληλο ταμείο μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καταπολεμήσει τον κοινωνικό αποκλεισμό. Χρειαζόμαστε μια ευέλικτη ισορροπία σε ό,τι αφορά τις θεματικές προτεραιότητες, ώστε το Κοινωνικό Ταμείο να μπορεί να κάνει περισσότερα για την κοινωνική ένταξη. Δεν μιλάμε εδώ για ποσά μόνο. Είμαι πεπισμένος ότι το θέμα είναι πώς θα χρησιμοποιηθούν τα ποσά αυτά, πώς θα χρησιμοποιηθούν καλύτερα, πώς θα σχεδιαστούν καλύτερα τα προγράμματα. Και αυτό απαιτεί μια πιο συμμετοχική προσέγγιση. Θα πρέπει και να σχεδιάσουμε καλύτερα τα προγράμματα, αλλά διάφορες περιοχές, διάφοροι, διάφορες μικροπεριφέρειες, διάφοροι δήμοι και κοινότητες έχουν διαφορετικές ανάγκες. Ε, άλλα, άλλες ανάγκες έχει ο Βορράς, ε, η Ονότος, η Αντολή, η μιας χώρας. Γι' αυτό έχει σημασία οι τοπικές αρχές και οι τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις να συμμετέχουν στο σχεδιασμό των προγραμμάτων αλλά και στην εφαρμογή τους. Τώρα, πώς θα προσδιορίσουμε τα ποσά. Τι ποσά χρειαζόμαστε. Αυτή τη στιγμή δημιουργηθούν ευρωπαϊκές πολιτικές. Είναι σημαντικό τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το, προφανώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να καθορίζει το ύψος των ποσών. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να αξιολογήσουμε σωστά τις ανάγκες προηγουμένως. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό οι εθνικές προτεραιότητες, οι τοπικές ανάγκες και οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες να συντονίζονται Uh, Φυσικά μπορούν να συνεχιστούν κάποιες άλλες επικαλύψεις. Μεταξύ των διαφορών ταμείων υπάρχει όμως ευελιξία. Δεν νομίζω ότι χρειάζομαστε περισσότερη ευελιξία, αλλά μεγαλύτερη σαφήνεια για να κατανοούμε καλύτερα τον ρόλο των ταμείων. Το Ταμείο παγκοσμιοποίηση. θέλω να το ενισχύσουμε, πρέπει, το έχουμε ανάγκη, αλλά πρέπει να βελτιωθεί η λειτουργία του. Καταλαβαίνω τις επικρίσεις και συμφωνώ ότι ο χρόνος που χρειαζόμαστε για να λάβουμε τις αποφάσεις είναι προβληματικός. Ε, συχνά όμως ε, ξαφνικά έχουμε μεγάλες απώλειες θέσεων ε, απασχόλησης και δεν υπάρχουν σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο πόροι για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Χρειαζόμαστε λοιπόν να συνεχίσουμε τη χρήση αυτού του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης. Με βάση την έκθεση θα ήθελα να συνεχίσουμε να βλέπουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία αυτού του ε, Ταμείου. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τώρα θα ακούσουμε τους ομιλητές. 1,5 με 2 λεπτά παρακαλώ. Βλέπετε όλοι, ο κύριος Επίτροπος χρειάζεται χρόνο για να απαντήσει και πρέπει να έχουμε και λίγο χρόνο εμείς για να ανακοινώσω και κάποια πραγματάκια για το τι θα γίνει με τις δικές μας εργασίες. Οπότε, Ανιέτ, όχι, Γιώραν Φέρμ τότε. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να ομολογήσω πως ανησυχώ λίγο για τη συζήτηση για το κοινωνικό ταμείο. Εάν δούμε τι έγινε με την πέμπτη έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αναφέρεται αυτό μόνο παρενθετικά. Εάν δούμε το τι γίνεται, επικεντρώνονται μόνο στα περιφερειακά ταμεία και τα περιφερειακά προβλήματα. Είναι σημαντικά. Μόνο παρενθετικά αναφέρεται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στην Σουηδική απάντηση εμεί μιλάμε για τις αραιοκατοικημένε περιοχές, σημαντικές, αλλά πολύ μικρότερο ποσοστό χρηματοδότηση από το Κοινωνικό Ταμείο που είναι πολύ μεγαλύτερο. Ένας λόγος είναι πως το Κοινωνικό Ταμείο και άλλοι ταμεί χρηματοδότηση δεν έχουν τους ε, ισχυρούς ε, δικαιούχου ε, που έχουν τα άλλα ταμεία. Δηλαδή περιφέρειες ε, με δημόσια χρηματοδότηση που χρηματοδοτούνται και από το Ταμείο για την ε, ε, ανάπτυξη κτλ. Ενώ άνεργοι μετανάστες κτλ. δεν μπορούν να ασκήσουν πίεση. Οπότε τι κάνει η Κομισιόν για να εξετάσει τα αποτελέσματα αυτά. Εγώ βλέπω λίγα πράγματα. Οπότε πρέπει να παλέψουμε για αυτό αν είναι να μην χάσουμε τη μάχη Δεύτερο και σύντομο. Ε, υπάρχουν δύο πτυχές ε, του Ταμείου. Να αναπτύξουμε δεξιότητες για αυτούς ε, που ήδη έχουν δουλειά και να βοηθήσουμε τους άνεργους ε, να εντάξουμε όσοι είναι μακριά από την αγορά εργασίας. Σε τι θα θέλετε να εστιαστείτε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Άλλα. Oui, merci, Madame le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και για τις πολύ ευγενικές σας ευχές. Σίγουρα τα γενέθλιά μου δεν θα μπορούσα να τα φανταστώ σε καλύτερο μέρος από ότι στην Επιτροπή σας με την δική σας παρέα. Λοιπόν, επανέρχομαι τώρα σε ένα πιο σοβαρό και πιο λυπηρό ζήτημα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, ακόμη και πριν από την κρίση, σε όλες τις χώρες μας διαπιστώσαμε μία αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας, ειδικά στους νέους, επιδείνωση της φτώχειας, μεγαλύτερη δυσκολία ένταξης κοινωνικής των μεταναστών, των αλλοδαπών. Οπότε στο μέλλον η απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου δεν μπορεί να είναι συνεχίζουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα, συνεχίστε να μου δίνετε τέτοια κονδύλια, θα συνεχίσω κι εγώ όπως πριν το έργο μου. Θα πρέπει να γίνουν αλλαγές. Τρεις παρατηρήσεις. Καταρχήν, στις περισσότερες χώρες, κανείς δεν ξέρει ότι υπάρχει ένα ταμείο που λέγεται Κοινωνικό Ταμείο. Κανείς δεν γνωρίζει ότι μερικά προγράμματα μόνο από το Κοινωνικό Ταμείο μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Είναι τεράστια η πρόκληση. Κάτι που θα αναφέρει φαντάζομαι η κυρία Ματέρα αργότερα και άλλοι. Το θέμα της διάκρισης μεταξύ του κοινωνικού ταμείου και αυτό που αποκαλούμε με πομπόδι τρόπο το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, θα πρέπει να γίνει η διαφορά αυτή σαφής. Είναι η ίδια φιλοσοφία, η ίδια πολιτική. Μπορούμε να έχουμε διαφορετικούς μηχανισμούς, αλλά δεν δικαιολογείται η ύπαρξη δύο διαφορετικών ταμείων για τον ίδιο στόχο. Θα πρέπει αυτή τη διάκριση κάπως να την εξετάσουμε. Επίσης, ε, η χρήση του Κοινωνικού Ταμείου και των άλλων διαθετικών ταμείων θα πρέπει να αφιερωθεί στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής του 2020. Σε ό,τι αφορά τους μείζονες κοινωνικούς στόχους της στρατηγικής του 2020, το ποσοστό δραστηριοποίησης των πρεσβυτέρων και των νέων, ο αριθμός των νέων που εγκαταλείπει τη φοιτηση πριν αποκτήσει πτυχίο, το κατόφλι της φτώχειας, όλα τα εθνικά προγράμματα προσαρμογής υστερούν σε σχέση με τους στόχους της στρατηγικής του 2020. Δεν θα πρέπει να γίνει κάποια ευθυγράμμιση και να πούμε θα εφοδιάσουμε με κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου τις χώρες που σέβονται στο, στα προγράμματά τους στην τήρηση των στόχων του 2020 για τους τομείς τους κοινωνικούς. Ευχαριστώ αλλά, ε, ξέρεις, σου έδωσε δώρο για τα γενέθλιά σου η Επιτροπή 36 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, Λαμπέρ. Και εγώ βεβαίως ε, εύχομαι τα χρόνια πολλά. Αλλά τώρα όσον αφορά τις επιλογές που έχουμε. Κοιτάξτε, λέτε πώς θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που έχουμε στην πολιτική αυτή και κάτω από αυτή την ομπρέλα βρίσκεται η περιφερειακή και εδαφική συνοχή. Αλλά στο σύνολο αυτό πρέπει να υπάρχει ευελιξία που υπάρχει εντός των κρατών μελών για να κάνουν κάτι περισσότερο όσον αφορά στο Περιφερειακό Ταμείο ή αν θεωρούν κάτι περισσότερο να δώσουν βάρος στο Κοινωνικό Ταμείο δεν μπορεί να μιλάμε για αποκεντρωμένη διοίκηση και να μειώνεται αυτή στο μέλλον. Δεν μιλάμε για, λίγο, για περισσότερη ευελιξία, να διατηρήσουμε αυτή την οποία που υπάρχει, κατόπιν. Ασχολήθηκα πάρα πολύ στη δεκαετία του 90 με τα κοινωνικά ταμεία και μετά πήγε στα Υπουργεία και στις περιφέρειες. Κοιτάξτε, εκεί πέρα έγινε ένα ξένο σώμα και θα πρέπει τελικά να πούμε πως η Ευρώπη 2020 δεν είναι κάτι θεωρητικό σε εθνικό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να συνδεθεί με αυτά τα οποία γίνονται για την εκπαίδευση των ανθρώπων, ανάπτυξη, την ανάπτυξη δυνατοτήτων και τη συμμετοχή στην πολιτική. Και θεωρώ πως κάποια κράτη-μέλη έχουν κάνει ε, λάθη νομίζω και θα πρέπει να κινητοποιηθούν καλύτερα. Ευχαριστώ. Κίνγκα Γκιόντς. Ευχαριστώ. Uh, θα ήθελα να συνεχίσω εκεί που σταμάτησε ο Γκόραν Φέρμ. Όταν μιλούμε για το κοινωνικό ταμείο, ανακύπτει το ερώτημα τι στήριξη μπορεί να έχει το ΕΚΤ. Και νομίζω ότι είναι και δική μας ευθύνη να δώσουμε αυτή την υποστήριξη στο κοινωνικό ταμείο. Επίσης έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις για τους Ρωμά. Αυτή τη στιγμή εκπονούμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ένταξη των Ρωμά με βάση την έκθεση της ειδική Ομάδας Εργασίας. Δεν έχουμε όμως πληροφορίες για το πώς βοήθησαν τα κονδύλια για τη βελτίωση της κατάστασης των Ρωμά, αν είχαν πρόσβαση οι Ρωμά στα κονδύλια αυτά. Το θέμα είναι να φτάνουν αυτά τα κονδύλια και στις ε, λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, στις μειονεκτούσες περιοχές και στους ε, ανθρώπους που πραγματικά τα χρειάζονται. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα, την καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε και την πολιτική, την πολιτική μας δέσμευση για να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτής της ε, ομάδας, των Ρωμά, σε όλη την Ευρώπη, γιατί η κατάστασή τους είναι δυσχερής όχι μόνο στις νέες χώρες μέλη αλλά και στις παλιές. Έχετε κάποια στοιχεία και ποιες είναι οι σκέψεις σας για να βελτιώσουμε την κατάσταση για την καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων. Μερικές φορές χρειάζονται και έκτακτες παρεμβάσεις. Πώς θα ε, βελτιώσουμε αυτή την προσέγγιση και τον τρόπο διαχείριση των κονδυλίων, ώστε να φτάνει και στου πληθυσμού Ρωμά. Κυρία Ματέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τον Επίτροπο που ήρθε εδώ και θέλω να επανέλθω στο πρώτο βήμα τη παρέμβασή του που μίλησε για τη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και ότι θα πρέπει αυτό να συνδεθεί με άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Θα ήθελα λοιπόν να, ακριβώς γι' αυτό να μιλήσω ε, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, που είπε ένα συνάδελφος προηγουμένως ότι αφορά, ενδιαφέρει πάρα πολύ το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να μας δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις. Το 2010 αυτό το ταμείο αποδείχθηκε ότι είναι πολύ χρήσιμο χάρη και στην πρικοδότηση του Ταμείου αυτού και χάρη στο διπλό στόχο του Ταμείου, δηλαδή για την οικονομική κρίση και για την ε, προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Μέσω μιας μεταρρύθμισης που έγινε και που την υποστήριξε το Κοινοβούλιο μέσω της έκθεσης πρωτοβουλίας ε, της, ε, του συναδέλφου Πόρτας, για τη σημασία βελτίωση τη λειτουργία αυτού του Ταμείου, ούτω ώστε να χρησιμοποιείται πιο γρήγορα και να χρησιμοποιείται και καλύτερα το Ταμείο, ε, πετύχαμε κάποια σημαντικά πράγματα. Λοιπόν, χωρί ε, πανηγυρικού και χωρί περικοκλάδε, θέλω να μου απαντήσετε απλά. Πιστεύετε σε αυτό το ταμείο, Πιστεύετε ότι πρέπει να συνεχιστεί μετά το 2013. Πιστεύετε ότι είναι συμπληρωματικό με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και κυρίως, πιστεύετε ότι μετά το 2013 αυτό το ταμείο ε, μπορεί να βοηθήσει στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης. Ο Ζωζέ Μανουέλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση που θεωρώ απλή και εύκολη. Και θα ήθελα να την ε, απευθύνω στο Επίτροπο. Το κοινωνικό ταμείο είναι συμμετοχικό. Ε, βοηθάει στην ανάπτυξη για όλους. βοηθάει σε μια έξυπνη ανάπτυξη, σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Τι θεωρεί ο Επίτροπος ότι είναι ανάπτυξη συμμετοχική, ανάπτυξη για όλους. Έπειτα, οι πέντε στόχοι της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Ειδικά αυτοί που είναι κοινωνικής φύσεως. Μιλήσαμε για το στόχο του 10% στις επενδύσεις, μιλήσαμε για την καταπολέμηση της ε, φτώχειας και για το στόχο του 20 για τα 20 εκατομμύρια. Μιλήσαμε για το 40% των νέων μεταξύ 30 και 34 ετών να αποκτήσουν ένα πανεπιστημιακό δίπλωμα. Αυτή είναι σημαντική στόχη. Το κοινωνικό ταμείο δεν θα πρέπει να είναι το ταμείο που θα έπρεπε να συμβάλλει για την υλοποίηση των στόχων αυτών δεν βλέπουμε ούτε στις α, ε, επίσημες θέσεις, ούτε στα έγγραφα να έχει τέτοια συμβολή το κοινωνικό ταμείο, ιδιαίτερα για την ένταξη των νέων στην κοινωνία. Φαίνεται ότι οι νέοι αποκλείονται και από τα έγγραφα και από τις ε, θέσεις τις επίσημες. Δυστυχώς ε, λείπει αυτή η πολύ σημαντική προσέγγιση από τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ και Μαρία Καρβάλιο. Ευχαριστώ. Συνεχίζοντας τη σκέψη του προλαλήσαντα, θα ήθελα να πω ότι μία εμπειρία που είχαμε στην Πορτογαλία είναι ότι οι δείκτες καινοτομία και προσόντων εξειδίκευση έχουν βελτιωθεί αισθητά χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είχαμε ένα πρόγραμμα χρήσης των κονδυλίων του Κοινωνικού Ταμείου για υποτροφίες ε, ανώτερης εκπαίδευσης και για διδακτορικό, μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό. Ε, επίσης, ε, είχαμε επιμόρφωση επιστημόνων που μετά συνέχισαν να, να απασχολούνται είτε στη δημόσια διοίκηση είτε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, σημαντικός εξυγχρονισμός των Δωμό στην Πορτογαλία έγινε χάρη στην συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ήταν πολύ θετική η εμπειρία μας λοιπόν από τη χρήση των κονδύλιων. Η χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου υπέρ της επιστήμης, ε, της έρευνας, της καινοτομίας τεχνολογικής ανάπτυξης, ε, χάρη στην ε, κατάλληλη συμμετοχή των νέων, δεν θα είναι ένας καλός τρόπος για την χρήση του Κοινωνικού Ταμείου στο νέο πλαίσιο το δημοσιονομικό. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επιτροπέ, έχετε τώρα την ευκαιρία να απαντήσετε στο δεύτερο γύρο των ερωτήσεων. Uh, uh, να ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησα, ε, απαντώντας για τα θέματα του Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση. Φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά κρεμή και ανοιχτά θέματα. Αλλά είναι και ξεχωριστό θέμα από το Κοινωνικό Ταμείο αυτό. Πιστεύω ότι ο λόγος που δεν πρέπει να συνεχιστεί το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης μετά 2013 δεν έχει να κάνει με την κρίση. Ε, το Ταμείο αυτό δεν δημιουργήθηκε ούτως ή άλλως για, ως απάντηση για την κρίση, αλλά πριν την κρίση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δυναμική οικονομία σημαίνει δυναμική αγορά εργασίας και σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο οι πολυεθνικές ε, οδηγούν, και η πολιτική των πολυεθνικών οδηγούν σε μείωση των θέσεων απασχόλησης. Οι κυβερνήσεις δεν έχουν τους πόρους να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις Και το πρόβλημα είναι ότι έχουμε ένα μακρό χρόνο μέσα στον οποίο παίρνουμε τις αποφάσεις, πρέπει να τον μειώσουμε. Ε, υπάρχουν πολλές συζητήσεις για την επιλεξιμότητα, υπάρχουν πολλές αφησιμίες ε, οι οποίες θα πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν. Αν λύσουμε αυτά τα θέματα θα υπάρξει πραγματική υποστήριξη. Εγώ πιστεύω ότι ιδανικά πρέπει να είναι χωριστό ταμείο. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες λύσεις για να κρατήσουμε τη λειτουργία. Το θέμα είναι να κρατήσουμε τη λειτουργία του ταμείου αυτού. Του ταμείου δηλαδή προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Θα επανέλθουμε όμως αυτό σε μεταγενέστερη φάση η Ευρώπη για το 2020 είναι το πλαίσιο από το οποίο ξεκινήσαμε και στο οποίο πάντα επιστρέφουμε. Καλωσορίζω τα σχόλια των συναδέλφων που λένε ότι πρέπει να υπάρχουν όροι ε, επιλεξιμότητας αυστηρή, ούτως ώστε οι χρήστες, οι τοπικές αρχές να ευθυγραμμίζουν τις πολιτικές τους και τα προγράμματά τους με τους στόχους της στρατηγικής 2020, ε, εστιάζοντας στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στη μείωση της στόχιας. Όλα αυτά τα πράγματα είναι αλληλένδετα και οι στόχοι της στρατηγικής 2020 είναι σοβαροί και είναι σχεδιασμένοι ούτως ώστε να είναι και φιλόδοξοι αλλά και ρεαλιστικοί. Και θα γίνουν και θα παραμείνουν ρεαλιστικοί αν έχουμε τα μέσα, τα εργαλεία για να υποστηρίξουμε την εφαρμογή τους. Πρέπει να εστιάσουμε στους τομείς εκείνους όπου υπάρχουν συγκεκριμένες προκλήσεις. Και τα προγράμματα πρέπει να είναι εστιασμένα επίσης. Ένα από τα παραδείγματα ε, ειδικού προγραμματισμού είναι η κατηγορία των Ρωμά. Είναι πολύ ψηλά στην, στις προτεραιότητές μας και λόγω του ότι είναι πολύ σημαντικό για την Ουγγρική Προεδρία. Το έχουμε συζητήσει με την Ουγγρική Προεδρία, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε περισσότερα κονδύλια για αυτούς. Ε, διάφορες κοινότητες περιθωριοποιημένες, όχι μόνο οι Ρωμά, αλλά και οι μετανάστες, δυσκολεύονται να καταλάβουν για ποιο λόγο υπάρχουν τα κοινοτικά ταμεία, πολλό δε μάλλον τα χρησιμοποιήσουν. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μια εδαφική προσέγγιση, δηλαδή να εντοπίζουμε τις μικροπεριοχές ή τις περιφέρειες, μικροπεριφέρειες ας πούμε, που πλήττονται περισσότερο. Χρειαζόμαστε καλό λογισμικό, ούτως ώστε να Προσαρμόζουμε δηλαδή τα ταμεία στο τοπικό πλαίσιο. Και λόγω της φύσης των προγραμμάτων χρειαζόμαστε και ιδέες για το πώς θα δώσουμε θέσεις απασχόλησης για αυτούς που έχουν λίγες δεξιότητες. Η κατάρτιση ήταν βασικό στόχος του Κοινωνικού Ταμείου. Αλλά λόγω των προβλημάτων και, του, και του κατεπήγοντος χαρακτήρα πρέπει να δώσουμε δουλειά σε ανθρώπους που δεν έχουν προσόντα. Και πρέπει να βοηθήσουμε τις ε, εθνικές κυβερνήσεις ε, σε αυτόν τον τομέα εφόσον θέλουν πραγματικά να προωθήσουν την κοινωνική συμμετοχή και ένταξη. Πρέπει να είμαστε σοβαροί για την ε, πολλαπλή συμμόρφωση την επιλεξιμότητα και τους όρους επιλεξιμότητας. Ε, πρέπει να τονίσουμε τους πολιτικούς στόχους και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να διατηρήσουμε σε κάθε γωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα κριτήριο επιλεξιμότητας. Δεν, δεν ισχύει ότι ξεκινάμε από το μηδέν, απλώς πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας καλύτερα και πρέπει να εργαστούμε πιο αποτελεσματικά με τους εταίρους μας, να εμπλέξουμε επίσης και τις κοινότητες που μας αφορούν. Ε, δηλαδή, όταν μιλάμε για τους ε, φτωχούς, θα πρέπει να εμπλέξουμε ε, στην προσπάθειά μας τους φτωχούς. Όταν μιλάμε για τους Ρωμά, θα πρέπει να εμπλέξουμε τις οργανώσεις των Ρωμά. Και θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία των τοπικών αρχών, των κυβερνήσεων, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των φορέων των κοινοτήτων αυτών. Αν μου δίνετε περισσότερο χρόνο, κυρία Πρόεδρε, θα συζητούσαμε περισσότερο και τα πολιτιστικά θέματα, γιατί συνδέονται αυτά με άλλε μεγάλες συζητήσει στην Ευρώπη. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για την ένταξη. Αλλά αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι το άνοιγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ε, διεύρυνση, στη μετανάστευση κτλ. έχει επιπτώσει στην αγορά εργασίας, έχει επιπτώσει στην εκπαίδευση και κυρίως στις ε, περιθωριοποιημένες κοινότητες, από όπου και αν προέρχονται. Το θέμα είναι καυτό για την Ευρώπη σήμερα. Και γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέου τύπου προγράμματα, νέες διευθετήσεις, νέες υποχρεώσεις. Δεν σημαίνει ότι όλα πρέπει να είναι καινούργια όμως. Ε, τελευταία χρονιά έκανα δύο ταξίδια στην Πορτογαλία. Είδα πράγματα που συνδέονται με τη σημερινή συζήτηση. Παραδείγματο χάρη για την επαγγελματική κατάρτιση. Ε, είδα πώς δημιουργούνται θέσεις, ας πούμε, για ανθρώπους με ειδικέ ανάγκες. Ε, πρέπει να εντάξουμε περισσότερους ανθρώπους με ειδικέ ανάγκες, είτε με μερική απασχόληση, είτε με πλήρη απασχόληση στην αγορά εργασίας. πρέπει όμως να έχουμε μια εστιασμένη προσέγγιση. Υπάρχουν παραδείγματα που μπορούν να μας εμπνεύσουν ιδίω για την επαγγελματική κατάρτιση, μέσω αυτής έχουμε ευκαιρίες να δώσουμε δουλειά σε ανέργους, αλλά και σε άλλου εργαζόμενους που βρίσκονται σε φάση μετάβασης και πρέπει να αναπτύξουν ε, προσόντα επίπεδου 21ου αιώνα. Είναι σε μεταβατική φάση γιατί ενδεχομένω περνάνε μια φάση ανεργίας. Ε, βέβαια υπάρχει και η διάσταση της αλληλεγγύη. Η εικόνα συμπληρώνεται μόνο όταν μιλήσουμε για αλληλεγγύη. Συμμετοχή όλων. Σημαίνει πιο δίκαιη η ευρωπαϊκή οικονομία. Ε, προσαρμογή του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου στον 21ο αιώνα και στις πραγματικότητες του, στις προκλήσεις μετά την εποχή της κρίσης. Μέσα σε μια παγκόσμια οικονομία όπου ο ανταγωνισμός είναι αβυσαλαίος, Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλους τους πόρους και τους ανθρώπινους πόρους. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε καμία κοινωνική ομάδα. Και η στρατηγική νομίζω του 2020 ε, δίνει ένα καλό πολιτικό πλαίσιο. Τώρα θα πρέπει να την εφαρμόσουμε με την κατάλληλη οικονομική υποστήριξη. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Kommissar. In der Tat. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Όντως, δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε ένα μόνο, ε, σε μία μόνο κοινωνική ομάδα και έτσι να το περιθωριοποιήσουμε. Και δεν είναι μόνο τα κράτη-μέλη που θα πρέπει να προσπαθήσουν να εντάξουν περισσότερο τις γυναίκες στην αγορά εργασίας. γιατί χρειαζόμαστε την πολύτιμη συνεισφορά και των γυναικών ε, για να τροφοδοτήσουμε την οικονομία μας και είναι κρίμα να στερούμαστε αυτή την πολύτιμη συμβολή. Ελπίζω, μια και όλοι συμφωνούμε, να βελτιωθεί η κατάσταση. Σαλβαδόρ, έχετε τον τελευταίο λόγο μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Επίτροπε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την υπεράσπιση του κοινωνικού ταμείου. Είναι ρόλος σας αυτός, το κάνετε πολύ καλά. Νομίζω ότι το ταμείο αυτό έχει τεράστια σημασία στο σημερινό δημοσιονομικό πλαίσιο και πρέπει να συνεχίσει να έχει παίζει αυτό το ρόλο για να πετύχει την οικονομική και κοινωνική συνοχή και την εδαφική συνοχή εκατομμύρια ανέργους έχουμε σε όλη την Ευρώπη και αυτοί αυτό ακριβώς ζητούν από το Κοινωνικό Ταμείο. Πέρα από τα θέματα επικουρικότητας, το Κοινωνικό Ταμείο έχει σημαντικό ρόλο και πρέπει να τον παίξει. Σημειώνουμε την άποψη του Επιτρόπου ότι, Επιτρόπου ότι αυτή η μείωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου από την περίοδο 90-93 στο 40% μέχρι σήμερα στο 20% δεν θα πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον. Το κοινωνικό ταμείο θα πρέπει να κρατήσει ε, τα ποσά του. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη δημιουργία συντονισμών, συνεργειών με τα διορθωτικά ταμεία, με το Περιφερειακό ταμείο, ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Γεωργικό Ταμείο, το Ταμείο Αλληλείας Όπως είπε και ο προηγούμενος επίτροπος, ο κύριος Χάν, θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική εστίαση ε, στον τρόπο διαχείρισης των ταμείων μέσω ενός κοινού στρατηγικού πλαισίου και μέσω ενός συντονισμού ε, των διαφόρων αρχών. Έτσι θα πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα αυτού του ταμείου που είναι θεμελιώδες για την πολιτική συνοχή στην Ευρώπη. Τονίζουμε επίσης, και το τόνισαν και διάφοροι συνάδελφοι, τη δυσκολία που έχουμε με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ε, ο τρόπος που εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη, ε, στις περιφέρειες και σε τοπικό επίπεδο, ε, καθιστά δύσκολη την εφαρμογή του. Και συχνά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ε, υπόκειται σε διαφορετικούς κανόνες. Οι Κομισιόν και οι υπηρεσίες της Κομισιόν ε, εφαρμόζουν διαφορετικούς κανόνες από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Ε, χρειάζεται πραγματικά μια πλούστευση αυτών των κανόνων. Ποιο είναι το μέλλον του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το είπαν ορισμένοι, συνάδελφοι, κυρίως η κυρία Ματέρα, και απάντησε ο Επίτροπος. Απάντησε ότι το Ταμείο αυτό παγκοσμιοποίησης θα πρέπει να συνεχίσει και μετά το 2013, αλλά παραμένουν κάποια ανοιχτά ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε. Θα πρέπει ένα τμήμα να χρηματοδοτηθεί ε, από ίδιους πόρους. Θα πρέπει να προσαρμοστεί στην παγκοσμιοποίηση ή θα το διατηρήσουμε ως ένα έκτακτο μηχανισμό ε, υπεράσπισης μας από την κρίση. Αυτά τα ερωτήματα ε, προκύπτουν από την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και θα πρέπει να επιληθούν στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. το ταμείο αυτό, ε, από ό,τι φαίνεται από τους διάφορους δείκτες των κρατών μελών, είναι ενδιαφέρον όργανο για το μέλλον. Φυσικά θα πρέπει να αποκτήσει και νέες ε, υποχρεώσεις στην κοινωνική ένταξη. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, όπως την ένταξη των Ρωμά. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αφορά δύο διαφορετικά πράγματα. Την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική. Εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την, τον άξονα της επικουρικότητας, αλλά είναι και κλειδί για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα μέσω της κατάρτισης των ανθρωπίνων πόρων. Γι' αυτό λοιπόν η συζήτηση που πρέπει να κάνουμε είναι αν θα πρέπει να το εντάξουμε στα, να έχει σαν στόχο μάλλον την έξυπνη ανάπτυξη ή την συμμετοχική ανάπτυξη. Ε, αυτό με σκοπό να υλοποιήσει τους στόχους στρατηγικής Ευρώπη 2020. Από την άλλη βέβαια θα πρέπει τα κράτη-μέλη να κρατήσουν την ευελιξία τους, ούτω ώστε να δημιουργήσουν το δικό τους μείγμα. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δηλαδή και Ευρωπαϊκό Ταμείο α, Περιφερειακής Ανάπτυξης η κατάσταση που υπάρχει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος διαφέρει, γι' αυτό χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία τη στιγμή προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αλλά και όχι μόνο, και των υπολείπων ταμείων. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν ε, ευρεία η συζήτηση και πολύ διεξοδική και όλα τα σχόλια που ακούσαμε στη διάρκειά της θα χρησιμεύσουν στο Σαλβατόρ για να συντάξει την έκθεσή του. Γιατί αυτό περιμένουμε από τον εισηγητή μας. Το Ταμείο Συνοχής, οι διαφορετικές πολιτικές, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο διαδραματίζουν νευραλγικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Σας ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ που είχατε την καλοσύνη να έρθετε στη συνεδρίες και ευχαριστούμε φυσικά και τον ε, κύριο Χάν, τον Επιτροπό Χάν που ήρθε νωρίτερα. Μου έχουν μείνει κάποιες ανακοινώσεις για το τέλος της συνεδρίασης. Στις 28 Φεβρουαρίου θα οργανώσουμε μία συνεδρίαση με θέμα τους πόρους, την κοινοτική χρηματοδότηση και τους κοινωνικούς πόρους. Γιατί υπάρχει ένα σύνδεσμος μεταξύ των ε, εσόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δαπανών της. Αυτό θα είναι το θέμα, τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θέμα της συνεδρίας της 28 Φεβρουαρίου. Θα μιλήσουμε και για τους ίδιους πόρους θα εξετάσουμε και κάποιους νέους ιδιοσπόρους. Ήδη οι συντονιστές ε, έχουν κάνει μία πρώτη διερεύνηση και πιστεύουμε ότι τα κριτήρια του νέου συστήματος ιδίων πόρων θα πρέπει να αναλυθούν. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αναπάντητα τα ερωτήματα της και τις απορίες των πολιτών και της Επιτροπής. Θα πρέπει να εξηγήσουμε ποιες είναι οι δικές μας επιθυμίες. Στην έκθεση αυτή θα μιλήσουμε και για τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν το σύστημα των ιδίων πόρων. Θα πρέπει άλλωστε να συζητήσουμε κατεπηγόντως και νέες μεθόδους, νέους τρόπους χρηματοδότησης. Και το πώς θα προσαρμόσουμε την κοινοτική μέθοδο σε αυτές τις νέες μορφές χρηματοδότησης. Η συζήτηση ακόμη και εκτός της Επιτροπής μας δείχνουν ότι η κοινοτική μέθοδο μερικέ φορέ γίνεται όμοιρο των συζητήσεων. Θα πρέπει όμω να διαφυλάξουμε αυτή την κοινοτική μέθοδο ακόμη και μετά τη θέση σε εφαρμογή τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Σημειώστε το λοιπόν, στι 28 Δευτέρου θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων και με τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι που είναι ο αρμόδιο καθήλυν για το θέμα αυτό και θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψει και με τον Φιλιπ Μέιστατ, τον πρόεδρο της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και μπορεί να μην έχει οριστικοποιηθεί πλήρως το πρόγραμμα, αλλά θα, θα σας το κοινοποιήσουμε μόλις αποσαφινιστεί. Λοιπόν, είχαμε επιτέλους ε, το τοκετό μετά από μια κοιοφορία αρκετά χρονοβόρα χθε και μάλιστα χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε και βριουλκό στο δοκετό. Ο τίτλος τη έκθεσης του Σαλβαντόρ θα είναι «Επενδύουμε στο μέλλον». Νέα, νέο δημοσιονομικό, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για μια ευφυή, ε, ανταγωνιστική και συμμετοχική Ευρώπη. Επιτέλους καταφέραμε και καταλήξαμε σε ένα τίτλο για την έκθεση της Επιτροπής μας. Καλά, βρήκαμε τον τίτλο. Χρειαζόμαστε όμως και ένα φύλλο πορείας για να δούμε πώς θα προσεγγίσουμε την κατάρτιση αυτής της έκθεσης. Εσείς έχετε λάβει αυτό το φύλλο πορείας, εγώ όχι όμως, ελπίζω να μην είναι κακός ιονός. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι έχουμε στην Επιτροπή μας αρκετό χρόνο για να καταθέσουμε τροπολογίες ως προς το σχέδιο έκθεση του Σαλβαντόρ Γκαρίγκα και θα προβλέψουμε αρκετό χρόνο και για τη συζήτηση. Θα συντάξουμε μάλιστα και συμβαστικές τροπολογίες. Υπάρχει χρόνος και για αυτές. Θα ήθελα λοιπόν να σας θέρμα παρακαλέσω αγαπητοί συνάδελφοι να ενημερώστε και τις πολιτικές σας ομάδες για, τη δραστηριότητα, για τις δραστηριότητές σας ώστε να λάβουν γνώση οι ομάδα σας το συντομότερο δυνατό των συζητήσεων εδώ. Στην 13η εβδομάδα, 21 Τρίτου, θα λήξει η διορία για την κατάθεση τροπολογιών. Μέχρι τότε θα πρέπει να είναι γνωστές οι θεμελιώδεις θέσεις των ομάδων. Και το αργότερο την 15η εβδομάδα θα πρέπει να είμαστε σε θέση να λάβουμε μια θέση επί της αρχής για τις συμβαστικές τροπολογίες. Νομίζω ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι αρκετά βολικό και ευελπιστούμε ότι θα υποβάλουμε την έκθεση στο Στρασβούργο τον Ιούνιο για να ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Και μάλιστα αν όλες οι ομάδες εργαστούν καλά και δώσουν εγκαίρως, εμπρόθεσμα, κοινοποιήσουν τη γνώμη τους, Είμαι σίγουρη ότι δεν θα έχουμε πληθώρα τροπολογιών στην Ολομέλη, γιατί αυτό πραγματικά θα ήταν ολέθριο. Γιατί πολύ συχνά είχαμε τέτοιο φαινόμενο σε εκθέσεις πρωτοβουλίες, μία πλημμυρίδα τροπολογιών 300 και στην Ολομέλεια, κάτι που θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθεί. Εγώ θα προσπαθήσω να αποφύγω τέτοια παρεκτροπή. Στις 10 Μαρτίου το πρόγραμμα εργασιών μας έχει ένα κενό. Δεν περιλαμβάνεται κανένα θέμα για τη 10 Μαρτίου. Είπαμε ότι στη συνεδρίαση αυτή θα μιλήσουμε για ό,τι μας έχει περισσεύσει, για όλα τα κρεμή ζητήματα. Συζητήσαμε το θέμα αυτό με τους συντονιστές Υπερβλήθησαν αρκετέ ιδέες και πολλές ιδέες είπαν ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το θέμα της χρηματοδότησης, της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Για να δούμε πώς εντάσσεται αυτή η προσπάθεια καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών στις υπόλοιπες μας δραστηριότητες. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό το θέμα να το συζητήσουμε. Και να δούμε και τις νέες αρμοδιότητες που αναλαμβάνουμε μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και έχουμε και κάποια διοικητικά θέματα αυτά των οργανισμών. Φυσικά δεν πρόκειται στη συνεδρία της 10 Μαρτίου να διεκπαιρεώσουμε όλους με κρεμότητες, αλλά θα έχουμε μια νέα ευκαιρία τον Απρίλιο να το κάνουμε και να προσαρμόσουμε αντίστοιχα και την έκθεσή μας. Αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε λάβει και τον κατάλογο με τις επιτροπές που έχουν ε, υποβάλει γνωμοδοτήσεις ή έχουν κοινοποιήσει τις θέσεις τους στην Επιτροπή μας. Δεν πρόκειται να σας διαβάσω ολόκληρο τον κατάλογο. Σε ό,τι φορά τώρα τα Εθνικά Κοινοβούλια, Μερικά κοινοβούλια μας έστειλαν τις απόψεις τους. Περιμένουμε και τις υπόλοιπες θέσεις των άλλων βουλών και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα είδος συμπίλησης αυτών των θέσεων. Αυτά. Άλλες ανακοινώσεις δεν έχω. Υπάρχει τίποτα στα διάφορα. Όχι. Πολύ ωραία. Καλό σας μεσημέρι και καλή σας όρεξη. Α, συγγνώμη, έχουμε και τούρτα γενεθλίων. Τούρτα γενεθλίων για τον Αλένα Μασούρ. Καλή όρεξη. Και καλό Σαββατοκύριακο, επειδή ευκαιρία. Ραντεβού στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα.